So, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. Έχω μια ενδιαφέρουσα ακρόαση. Έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Έχουμε ένα εξαιρετικό πάνελ για να συζητήσουμε για την σχετική μεταρρύθμιση. Ο κύριος Βίλεμ Παλενίκ, ο οποίος είναι μέλος τη Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Έχουμε τον κύριο Ζίγκφριντ Τζάξ, ο οποίο είναι επικεφαλή τη προστασία. τον δόκτωρο Στέφαν Χοχ Ράινα Στίγκλερ, ο οποίο ασχολείται με την πολιτική αντιμετώπιση των κινδύνων, τις ε, ε, των ευάλωτων καταστάσεων από το Ίδρυμα για την ανάλυση εφαρμοσμένων συστημάτων, τον κύριο Ντάντζελο, ο οποίος είναι επικεφαλής ε, της, προστασίας, ε, πολιτικής προστασίας του σχετικού τμήματος ε, της Ιταλικής κυβέρνησης και πρώτα πρώτα να δώσουμε το λόγο εις τον κύριο ε, Πάλενικ. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τώρα, να σας πω πρώτα πρώτα πώς βλέπει τα πράγματα η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή η οποία εκπροσωπεί τις οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών και επίσης έχουμε εκπονήσει μια γνωμοδότηση με την ομάδα εργασίας εγώ έχω συμμετασχεί εκεί και τον ε, Δεκέμβριο του 2013 εγκρίναμε αυτή την έκθεση αυτό το κείμενο. Η πρόταση της ε, Επιτροπής βασίζεται στην εμπειρία τη σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ταμείο Ελληνικής, κάτι το οποίο συμμετείχε το 2002 και αφορά τις φυσικές καταστροφές, τις θεομηνίες πρικοδότηση είναι ένα δισεύρα και εστιάζει την προσοχή του αυτός ή στην ε, κάλυψη αυτών των ε, καταστροφών και την ε, ανασυγκρότηση των περιοχών που τους εφίστανται. Η πρόταση αυτής της επιτροπης Επιτροπής πρώτα-πρώτα προσέχει αυτό το Ταμείο στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αυτό αφορά και κάποιες ε, καταστροφές ε, οι οποίες έχουν προκληθεί από φυσικά πρόσωπα. Σε σχέση με αυτή την πρόταση τώρα, δεν μπορούμε να πούμε γενικά, ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, τροποποίηση αυτού του κανονισμού. Επίσης, συμφωνούμε ότι χρειάζεται να μειωθεί η γραφειοκρατία ε, σε σχέση με την διαχείριση αυτού του ταμείου. Εμείς θέλουμε να υπάρξει μια πρικοδότηση, να υπάρχουν ε, καλύτερες συνθήκες και περισσότερη διαφάνεια. Αυτό ισχύει και με την κλιματική αλλαγή, η την καινούργια κατάσταση, η οποία αφορά τις φυσικές καταστροφές που θα χτυπήσουν και άρα χρειάζεται αυτό το Ταμείο η Ευρωπαϊκή Ένωση από δική μας πλευράς. Κάτι γνώμη μας. Η προθεσμία προβλέπεται για την εκταμείευση είναι πάρα πολύ μακρά σε σχέση με τι ανάγκε αυτού νου που έχει χτυπηθεί από την ε, καταστροφή. Ε, Επίση, εμεί αυτό το οποίο προτείνουμε σχετίζεται και με την κατάσταση τη της, της, σχετικής ε, περιφέρειας, σε σχέση με την κατασκευή κάποιο δάσο, όποτε θέλουμε να γίνει ένα δάσο ε, ε, δαπάνες αυτού του ταμείου και επίσης ε, θα πρέπει να προβλέπεται αυτή η αναδάσωση, κάτι το οποίο προσπαθούμε δεν προβλέπεται. Οπότε εμεί αυτό συγκεκριμένα προτείνουμε κάτι άλλο. Επίση το οποίο προτείνεται είναι το τι θα, πώς θα εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών όπως ο Ερυθρό Σταυρό έχει ρόλο να διαδραματίσει κοινωνία των πολιτών. Οπότε θα πρέπει να συμμετάσχει και να εμπλέκει με διαφορετικού τρόπου. Κάτι άλλο το οποίο τώρα προτείνει η Επιτροπή μα είναι το πώ θα έχουμε αντί για 1% του ΑΕΠ ε, σαν κάλυψη ε, γιατί θεωρούμε το 5% το πρώτο Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ε, υψηλό. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Δίνω τον λόγο στον κύριο Ζίκφριτ Ζάξο. I'm happy to share with you Με ιδιαίτερη χαρά να συμμεριστώ απόψε κάποιες από τις ε, εμπειρίες μου, τα βιώματά μου όσον αφορά την ε, λειτουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης στην Αυστρία, Ευρωπαϊκού Ταμείου από το 2012, 2002 ε, μέχρι σήμερα. Παρουσιάζω την προσέγγιση μιας αρχής που εφαρμόζει και λειτουργεί από ένα κράτος που ωφελείται από τις δράσεις αυτές και σε σχέση με αυτό υπάρχουν και κάποιες προσδοκίες. Το Ταμείο πρέπει να πετυχαίνει κάποιους γενικότερους στόχους, να εκφράζει, να είναι ένα μέσο αλληλεγγύης ε, για ειδικά γεγονότα. Πρέπει να μπορεί να κινητοποιεί επαρκή χρηματοδοτική βοήθεια έγκαιρα πρέπει να έχει εφικτές διαδικασίες, λειτουργικές διαδικασίες που θα στοχεύουν στο να αντιμετωπιστεί μια καταστροφή το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατικού χαρακτήρα με σαφείς κανόνες και κανονισμούς, με ελαστικότητα υλοποίησης και εφαρμογής, διαφάνεια, λογοδοσία. Όλα αυτά πρέπει να τηρούνται. Και θα πρέπει να είναι ένα μέσο το οποίο θα έχει ευδιάκριτο χαρακτήρα για τους πολίτες και θα είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό για τις εθνικές και περιφερειακές αρχές. Τα ζητήματα, τα θέματα που θα ήθελα να αντιμετωπίσω, δηλαδή πώς, ποιες επιδόσεις είχε το Ταμείο για να αντιμετωπίσει αυτές τις απαιτήσεις στην πρακτική εφαρμογή μέχρι σήμερα, θα ήθελα να επικεντρωθώ σε πέντε κύριες αρχές, πέντε άξονες. Ποιες διαδικασίες λειτουργούν σήμερα υπό τον κανονισμό του, του Ταμείου που θα έπρεπε ίσως να βελτιωθούν. Ποιοι κανόνες και κανονισμοί θα έπρεπε να βελτιωθούν. Ποιε είναι οι προσδοκίε των θυμάτων ή των τελικών αποδεκτών που επωφελούνται από αυτά τα κονδύλια. Μπορεί, μπορούν αυτά τα μέσα να λειτουργήσουν άμεσα και να φτάσουν στους δικαιούχους χωρίς γραφειοκρατική επιβάρηση. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα, δηλαδή πρέπει και να υπάρξει και απλούστευση κανόνων. Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ουσιαστικά είναι το ότι το Ταμείο καταρχήν λειτουργήσε με τρόπο αποτελεσματικό ήταν εφικτές και λειτουργικές οι δράσεις και η χρηματοδότηση από το Ταμείο, όμως τα διοικητικά βάρη, γραφειοκρατικά βάρη είναι υψηλά και θα πρέπει έτσι να τροποποιηθούν οι διαργασίες, οι διαδικασίες και να αποσαφινιστούν οι κανόνες. Η πρόταση για ένα νέο κανονισμό θεωρώ ότι βαίνει προς την ορθή κατεύθυνση και θέτει τα σωστά προβλήματα τα οποία θέλει να αντιμετωπίσει. Όμως από την άλλη πλευρά ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει υπερβολικό νέο βάρος ε, που θα δημιουργηθεί όσον αφορά την εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων και θα πρέπει να προσαρμοστούμε να είμαστε σε τεχνικό επίπεδο αποτελεσματικοί. Σε σχέση με τα μέχρι σήμερα θέλω να πω ότι η εφαρμογή όσον αφορά τα αιτήματα, τις αιτήσει η εφαρμογή και η υλοποίηση είναι το πιο κέριο θέμα. Τεχνικά εργαλεία ή μέσα που παρέχονται βοηθούν και βοήθησαν τις αρχές να κάνουν ε, σωστά τη δουλειά τους όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων και οι επεξηγήσεις που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μέχρι σήμερα πολύ επικοδομητικές. Συνολικά τώρα το χρονοπλαίσιο για, τον, για το Ταμείο, 10 εβδομάδες δηλαδή για το αίτημα το οποίο πρέπει να τεθεί, ένας χρόνος και έξι μήνες για την λειτουργία και ε, ανάληψη δράσης είναι ε, αρκετέ προκλήσεις, ωστόσο όμως θα πρέπει να δούμε και κάποια τροποποίηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί και κάποια απλούστευση θα μπορούσε να λειτουργήσει. Θα επανέλθω σε αυτό άμεσα στη συνέχεια. Η περίοδος εφαρμογής περίοδου διετούς φτάνει, ε, χρειάζεται ένα χρόνο για να φτάσουν τα χρήματα και μετά οι διαδικασίες μπορεί να θεωρηθούν χρονοβόρες. Ε, θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες και έτσι και μια παράταση, μια επέκταση θα μπορούσε να είναι ε, θετικό πράγμα. Δύο χρόνια δηλαδή από τη στιγμή κατά την οποία προκαλούνται οι πρώτες ζημιές. Είναι επαρκές χρονικό διάστημα νομίζω εγώ αυτό και να υπάρχει μία ενιαία πληρωμή σε σχέση με τις δράσεις, τα, περιορίζεται φυσικά σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες, δεν υπάρχει ανάγκη συγχρηματοδότησης και δεν χρειάζονται ενδιάμεσες εκθέσεις. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν επαρκής ε, ε, ευελαστικότητα για τα κράτη-μέλη να επιλέγουν τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και να, να επιλέγεται και ο κύκλος ε, των όσων θα ωφεληθούν θετική υποστήριξη και συμβουλέ δόθηκαν από τι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτέ είναι οι πτυχέ ε, που προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μέχρι σήμερα. Αυτό που θα μπορούσε να αναπτυχθεί είναι το οτιδήποτε θα βοηθούσε στι αιτήσει ε, που πρέπει να υποβάλλονται για την εκτίμηση ζημιών. Περαιτέρω οδηγίε κατευθυντήριε γραμμέ θα ήταν κάτι επωφελές αν μπορούσε να γίνει. Σύντομα, κάποιε τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειε θα ήθελα να αναφέρω για να καταδείξω τι εννοώ πάντα στις συζητήσεις διαδραμάτιζε ένα ρόλο το τι είναι η ζημιά. Άμεσα ή έμεσα κόστη θα πρέπει να καλύπτονται από το Ταμείο. Υπήρξε ήδη η διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το θέμα, σε σχέση με το ότι θα πρέπει να δούμε αν θα συμπεριλαμβάνεται ε, το ΦΠΑ ή όχι και αν θα υπάρχει αποκατάσταση, πλήρης αποκατάσταση σε σχέση με τις υποδομές άμεσης, άμεσου χαρακτήρα που πρέπει και αυτό να αποσαφηνίζεται, οι απώλειες σε σχέση με τα κόστη για την ανοικοδόμηση και ποιες είναι ακριβώς, ποιο είναι το εύρος των ζημιών κόστος ε, για τις απώλειες ή και κόστος και για τις υποδομές επιπλέον. Η διαφοροποίηση μεταξύ δημόσιων κρατικών ζημιών και ιδιωτικών ε, βλαβών ή ζημιών είναι και κάτι άλλο το μπορούσε να, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια περαιτέρω διαφοροποίηση. Επίσης, η εκτίμηση των ζημιών, ε, καθώς επίσης και το ποιες κατηγορίες θα μπορούσαν να εντάσσονται. Όσο πιο σαφείς είναι οι κανόνες και οι διατάξεις, τόσο καλύτερο θα είναι και επικοδομητικό για τους ε, όσους θα ωφεληθούν από αυτές τις δράσεις. Κάποιες κατευθυντήρες γραμμές είναι λοιπόν αναγκαίες για να είναι λειτουργικά τα κονδύλια αυτού του Ταμείου και να υποφελούνται οι αποδέκτες από αυτά τα χρήματα. Θα ήθελα τώρα να επιστήσω την προσοχή σας στα γυτνιάζοντα κριτήρια, γειτονικά κριτήρια που εφαρμόζονται μόνο με, σε χώρες με άμεσα σύνορα, με σύνορα σε σχέση με χώρες που έχουν υποστεί τέτοια πλήγματα. Και αυτό θα μπορούσε επίσης να εξετάζεται αν δικαιολογείται ή όχι, αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις ε, σε σχέση με αυτό το κριτήριο ως γνώμονα. Και μετά προφανές είναι ο έγκαιρος χαρακτήρας χορήγησης ε, της βοήθειας. Πρέπει να επιταχύνονται οι διαδικασίες λήψης απόφασης ε, ώστε η συνεισφορά με τα κονδύλια από αυτό το ταμείο προς τους ε, όσους έχουν ανάγκη, προκαταβολές για παράδειγμα, διάθεση χρημάτων άμεσα είναι κέρια σημασία στοιχείο. Τελευταίο, η έκθεση η υλοποίηση ή εφαρμογής Κάπως επιβαρύνεται και αυτό ο στοιχείο με γραφειοκρατικά εμπόδια. Υπάρχουν κάποια κρυφά ή συγκαλυμμένα γραφειοκρατικά εμπόδια όπως ε, σε σχέση με το πρότυπο συμφωνίας εφαρμογής που θα μπορούσε να απλουστευτεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται τα πράγματα για όσους ε, θα είναι αποδέκτες και θα ωφεληθούν από αυτά τα κονδύλια. Καθώς ερχόμαστε τώρα στην χρήση των κονδυλίων για τα θύματα ή τους αποδέκτες ε, Δηλαδή τι αναμένουν, τι προσδοκούν από το Ταμείο αυτά τα άτομα και ποια προβλήματα θα, μπορούν να, θα μπορούσαν να αντιμετωπίζουν. Ένα πράγμα είναι το πιο σημαντικό ίσως εδώ αποκατάσταση μετά από μια τέτοια θεομηνία, μετά από μια τέτοια καταστροφή είναι ανάγκη να αναλαμβάνεται άμεσα ως δράση και η βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης ε, πολλές φορές καθυστερεί. Λοιπόν, οι δράσεις ε, θα πρέπει να ξεκινούν και να γνωρίζουν ε, οι εποφελούμενοι ποιες είναι οι διαδικασίες σε σχέση με διαδικασίες που απαιτούνται από το Ταμείο. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται, χρειάζονται αυτά τα χρήματα και σε υστερότερο διάστημα. Οι διαδικασίες όμως των κρατών μελών ευθύς εξ αρχής πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις και διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης. Τα προβλήματα, οι τριβές που υπάρχουν πρέπει να αντιμετωπίζονται. Επιπλέον πρόσθετη έλεγχη σε σχέση με τις ε, εφαρμογές ε, προς όφελος των αποδεκτών προκαλούν και πρόσθετο έργο που πρέπει να καλύπτεται. Το πιο σημαντικό όμως θέμα ίσως είναι το ζήτημα Αυτά τα μέσα για τις χρηματοδοτικές, χρηματοοικονομικές ε, παρεμβάσεις φτάνουν γοργά, έγκαιρα σε αυτούς που τα χρειάζονται ή υπάρχουν ε, γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Υπάρχουν προτάσεις λοιπόν ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα μέσω προκαταβολών που θα καταβάλλονται. Υπάρχει ανάγκη να πλουστευτούν οι κανόνες. Μάλιστα ναι, αυτό είναι ήδη σαφές από προηγούμενες παρατηρήσεις και επεξηγήσεις. Απλούστευση λοιπόν τυποποίηση και μέσα σε ένα πλαίσιο τυποποίησης είναι αναγκαίο να λυθούν υπόψη κάποιες τεχνικές πτυχές. Δηλαδή ένα έγγραφο προς ανατολισμόν για ε, το πλήρες μέτρο και εύρος παρέμβασης που θα ήταν καλοδεχούμενο μέσα όπως πρότυπα ε, εντύπων ή εγγράφων που πρέπει να συμπληρώνονται θα ήταν χρήσιμα και αυτά. Δηλαδή και να υπάρχει και ένα πρότυπο έκθεσης που θα υποβάλλεται. Ουσιαστικά έχουν γίνει και έχουν καταδειχθεί αυτά από ένα μακρό κατά, μακρύ κατάλογο για τις παρεμβάσεις. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να επιταχυθούν οι διαδικασίες και να πλουστευτούν επιπλέον. Και ελπίζω ότι ήδη έχουν βρεθεί και έχουν υλοποιηθεί κάποιες εύθετες ε, αποτελεσματικές λύσεις που εντάσσονται και εμπεριέχονται σε μια πρόταση για κανονισμό που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Τώρα ευχαριστώ. Ε, thank you. Ε, ευχαριστώ. Ε, δόκτωρ Στέφαν Κοχράινεν Στίγκλερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η δική μου ομιλία αφορά ουσιαστικά κάτι που δεν έχουμε σε έγγραφο. Δεν ε, βλέπουμε τις πραγματικές υποκείμενες ανάγκες για τις φυσικές καταστροφές. Είναι κάτι που μπορούμε να διαχειριστούμε αξιολογώντας τους κινδύνους. Βασίστε σε πιθανότητε, ε, Εάν δεν ενσωματώσουμε αυτούς του κινδύνου, ουσιαστικά καταλήγουμε σε λάθο συμπεράσματα. Και εδώ ήθελα να κάνω μια παρουσίαση που αφορά αυτά τα ζητήματα των τριών διαστάσεων, τη στιβαρότητα του Ταμείου Αλληλεγγύη, την ε, νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα. Όπως ακούσαμε ήδη, το Ταμείο αλληλεγγύη υπάρχει ώστε να παρέχει αλληλεγγύη. Τι εννοούμε με την αλληλεγγύη, να βοηθάμε ανθρώπους σε κράτη όπου δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές διότι υπερβαίνουν την ικανότητα του κράτους. Ακούσαμε ήδη πώς αυτό έχει διαρθρωθεί. Έχουμε κονδύλια ενό δισεκατομμυρίου. Έχουμε αυτή την προσέγγιση με ένα κατόφλιο. Τα ακούσαμε όλα. Το επόμενο που πρέπει να συζητηθεί στη μεταρρύθμιση τώρα ουσιαστικά θέλω να συμπεράνω ότι να ξέρουμε ότι είναι αδύνατο να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιηθεί, έτσι λένε, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχει δυνατότητα αξιολόγηση του κινδύνου αυτού. Θέλω να σα δείξω εδώ πώς μπορεί να το αξιολογήσει κανεί, να το εκτιμήσει εκ των προτέρων και τι σημαίνει η αξιολόγηση των κινδύνων. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι όταν μιλάμε για ταμείο αλληλεγγύης, αυτό προτείνεται εδώ, είναι ότι θα πρέπει να έχει διερθρωθεί ως μηχανισμός κινδύνων. Πρέπει δηλαδή να αξιολογήσει κανείς την πιθανότητα να συμβούν εθνικές καταστροφές ε, ή φυσικές καταστροφές στις χώρες. Κάνοντας αυτό πρέπει να σκεφτεί κανείς ε, τη στιβαρότητα και τις υπόλοιπε διαστάσεις πιο λεπτομερώς. Βρίσκονται ενδεχομένω κάποιες λύσεις για προβλήματα που έχουμε αυτή τη στιγμή με το Ταμείο χρησιμοποιώντα αυτή την οπτική γωνία. Το πρώτο είναι ότι ένα από τα κύρια προβλήματα από την άποψη τη στιβαρότητας ε, ε, ας πάρουμε τις πλημμύρες. Οι πλημμύρε ε, είναι συνήθω μεγάλη κλίμακα, ε, έχουν μεγάλη κλίμακα επιπτώσει και συμβαίνουν συνήθω σε πολλέ χώρε ταυτόχρονα. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό οδήγησε στη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύα το 2002. Πολλέ χώρε αποτέλεσαν το αντικείμενο τέτοιων πλημμυρών παρατηρούμε αύξησή τους. Πρόκειται για τις ε, κύριες καταστροφές, ε, φυσικές καταστροφές, οφείλονται στην ε, κλιματική αλλαγή και σε άλλα, αλλά οι κλιματικές, κλιματικές προέλευσης καταστροφές αποτελούν το κλειδί ουσιαστικά του Ταμείου και τώρα αυτά, τα συμβάντα μεγάλης κλίμακας είναι εξαιρετικά δύσκολα και πιέζουν ιδιαίτερα το Ταμείο Ελεγγύης Πώς να τα αξιολογήσουμε. Πρώτον πρέπει να δούμε από τι Εδώ μπορείτε να δείτε το κόκκινο χρώμα δείχνει περιοχές ε, όπου αν συμβεί η πλημμύρα επηρεάζονται και άλλες περιοχές. Οι πλημμύρες λοιπόν ε, είναι συσχετισμένες, ειδικότερα υπό ακραίες συνθήκες. Και το Ταμείο Ελεγγύης ουσιαστικά αφορά ακραίες καταστάσεις για να βοηθήσει τον κόσμο να τις αντιμετωπίσει. Αυτές οι ακραίες καταστάσεις είναι που μας ενδιαφέρουν. Πώς θα το αξιολογήσει κανείς όσον αφορά την επικινδυνότητα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, αλλά θεωρητικά αξιολογεί κανείς τον κίνδυνο ώστε η κατανομή απολειών, ουσιαστικά η πιθανότητα να υπάρξουν απώλειες, ζημίες ε, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτιμώνται για κάθε μία από τις χώρες ε, με εφαρμογή των κριτηρίων κατοφλίου και έτσι έχει κανείς την κατανομή επικινδυνότητας για το Ταμείο Ελληνικής. Για ποιο λόγο, διότι έτσι μπορεί κανείς να αξιολογήσει την πιθανότητα οι αξιώσεις πληρωμών ε, κατά πόσο θα είναι υψηλότερε από το 1 δισεκατομμύριο και ουσιαστικά μπορεί να δει κανεί βάσει μια τέτοια ανάλυση ότι το Ταμείο Ελεγγύη επιδίδεται σε τέτοιε. ουσιαστικά αφορά τέτοιε μεγάλου ε, μεγέθου καταστροφέ. Κάθε 12 χρόνια περίπου μπορεί να είναι τόσο μεγάλε καταστροφέ που να υπάρξει υπέρβαση του κατοφλίου αυτού. Συμπεραίνουμε λοιπόν πρώτον ότι ακόμα και αν αυξήσουμε αυτό το Ταμείο είτε αυξάνουμε αυτό το ταμείο ενσωματώνοντας αυτές τις ε, μεγάλες καταστροφές. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες χρήση αυτού του ταμείου, αλλά όπως φαίνεται η δυνατότητα ανταπόκρισης του, το robustness όπως λέει ο μελίτης, ε, μπορεί να αυξηθεί ε, εάν έχουμε καταστάσεις που υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο, το κατόφλιο αυτό. Το επόμενο είναι το θέμα της ελληνικής. Πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουμε ικανότητες να ανταποκριθούμε. Εάν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια καταστροφή, τότε ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε βοήθεια εξωτερική. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βάσει κάποιων μοντέλων επικινδυνότητας, ε, δείτε το παράδειγμα της Αυστρίας, το οποίο φυσικά δεν είναι απόλυτο, το κατόφλιο για την Αυστρία είναι τέτοιο που όταν θα βοηθούσε το Ταμείο Λιλεγγύης στην Αυστρία θα έπρεπε ουσιαστικά να δώσει προτεραιότητα στην Ουγγαρία και την ε, ε, και τι δίπλα χώρες γιατί έχουν λιγότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να συσχετιστεί με την οικονομική απόδοση ή άλλα μέτρα. Actually, uh, would increase actually the, the... Έτσι λοιπόν οι χώρε μικρότερου εισοδήματο θα είχαν περισσότερο πλεονέκτημα στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύη. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για αλληλεγγύη ότι όλοι βοηθούν ε, όλου. Ουσιαστικά λαμβάνουν βοήθεια αυτοί που πραγματικά τη χρειάζονται. Η τελευταία διάσταση, η διάσταση τη απόδοση. Πολλέ φορέ συζητάμε για το πώ μπορούμε να μειώσουμε την επικίνδυνοτητα για το μέλλον. Πολλέ βελτιώσει έχουν επιτευχθεί. με την οδηγία για τις πλήμμυρες. Ε, εάν η μόνη απέτηση είναι ε, μια χαρτογράφηση του κινδύνου πλημμυρών, ε, δεν αρκεί για να μειωθεί ο κίνδυνος. Τι άλλο λοιπόν μπορούμε να κάνουμε, εάν τιμολογήσουμε τον κίνδυνο, μπορούμε να ορίσουμε πότε θα τον μειώνουμε και με ποια τιμή. Κατανέμοντας ουσιαστικά την επικίνδυνοτητα, κατακαιρματίζοντας την. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόσθετο ασφαλιστικό μηχανισμό όπου θα μειώναμε ε, την επικίνδυνοτητα μειώνοντας την τιμή της επικίνδυνοτητας. Assets uh, Ας δούμε ας πούμε τι έχει γίνει στο Μεξικό αλλά και σε άλλες χώρες ε, όπου τέτοιοι κίνδυνοι δεν θεωρούνται μη ασφαλιζόμενοι, μπορούν να αποτελεστούν αντικείμενο ασφάλισης. Ένα δεχόμενο λοιπόν θα ήταν ε, να τιμολογήσουμε ε, την επικίνδυνοτητα για αυτά τα δημόσια αγαθά και αν μειώσουμε τον κίνδυνο πρέπει να πληρώσουμε λιγότερα για να τον αποκαταστήσουμε. Αυτά τα τρία πράγματα θα ήθελα να πω το τελευταίο είναι τι μπορεί να κάνει εδώ το Ταμείο Εάν μπορεί κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσει αυτές τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, μπορεί να χρηματοδοτήσει κομμάτι αυτών των ε, ασφάλιστρων ε, για να είναι πιο φθηνές για τους φτωχότερους. Μπορεί επίσης να εξετάσει τους υψηλούς κινδύνους για κάποιες χώρες. Πολλέ ε, ασφαλιστικέ εταιρείε δεν δέχονται τόσο υψηλού κινδύνου στο χαρτοφυλακία του γιατί του κοστίζει πολύ. Έχουμε κάποιε περιπτώσει όπω στη Γαλλία όπου αυτοί οι υψηλοί κίνδυνοι αναλαμβάνονται από την κυβέρνηση ή άλλου μηχανισμού. Από το δημόσιο ουσιαστικά ή από κάποιον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Όλα αυτά τα πράγματα προσφέρουν αυτά τα ωφέλη ότι μπορεί κανείς να μειώσει τον κίνδυνο μειώνοντας τα χρήματα ε, που πρέπει να καταβάλει σε μια ασφάλεια. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι δυνατή διαφοροποίηση του κινδύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του μεγέθους της. Μια τέτοια διαφοροποίηση καθιστά πιο φθηνή αυτή την ασφάλιση και τις σχετικές συμφωνίες αντί να σκεφτεί κανείς ε, χώρα προς χώρα. Για να συνοψίσω, θα έλεγε κανείς ότι επινάψε η επικινδυνότητας ε, δεν βασίζεται σε απόλυτες τιμές ε, αλλά σε τιμές που επηρεάζουν τις επιδόσεις, την ε, δυνατότητα οικονομικής αντιμετώπισης που έχει μια χώρα. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί να αυξήσει τα κονδύλια του Ταμείου για να αυξήσει τη δυνατότητα αποκρισής του ή να παρεκτρέψει κάποια τέτοια κονδύλια στην ε, αγορά των ασφαλιών και μια άλλη δυνατότητα είναι να επαναπροσωτολίσουμε αυτό το Ταμείο Ελληνικής από ένα ταμείο που αντιμετωπίζει τα πράγματα μετά την καταστροφή σε ένα μηχανισμό που ε, ε, αντιμετωπίζει με τα κεφάλαια του προληπτικά τις καταστάσεις πριν επέλθουν οι καταστροφές μέσω συγκεκριμένων μηχανισμών. That's basically it. Thank you very much. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Thanks, thanks a lot. Ε, Mr. Luigi. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λουίτζι D'Angelo. έχετε το λόγο. Grazie, signor Presidente. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ανήκω στην Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ιταλίας. Πρόκειται για την αρχή η οποία συντονίζει τη χρήση αυτών των κονδυλίων στην Ιταλία συμμετέχοντας συνεργατικά μαζί με άλλες διοικήσεις που το υλοποιούν όπως για παράδειγμα οι περιφέρειες. Εγώ ανήκω σε μια χώρα που έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν ε, τη μισό από όλα τα κονδυλία που έχουν δοθεί από το 2002 μέχρι σήμερα. Για εμάς φυσικά ήταν πολύ σημαντικός αυτός ο μηχανισμός όπως καταλαβαίνετε Αναγκαίως μάλιστα διότι μας έπληξαν ε, σημαντικές καταστροφές που γνωρίζουν όλοι. Από μια άποψη λοιπόν εμείς ήμασταν ουσιαστικά και το πεδίο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε περισσότερο αυτό το ταμείο ε, κατά επανάληψη υπό πολύ διαφορετικές ε, περιστάσεις και υπό πολλές διαφορετικές περιστάσεις μας και επικρίσεις αλλά πιστεύω ότι για μας ε, είναι μεγάλη ελπίδα αυτός ο νέος ο κανονισμός γιατί για μας οι διάφορες εφαρμογές ε, του ταμείου αυτού ε, συμβάλλουν σε αυτό το νέο κανονισμό. Χρειάζεται πιστεύουμε αυτή την αναθεώρηση. Αυτό που θέλω να πω αμέσω είναι το εξή. Κατά την άποψή μα, το Ταμείο Ελληνική, τουλάχιστον όσον αφορά τα όσα έχουν συμβεί στην Ιταλία, αύξησε πολύ σημαντικά την ε, συνείδηση ότι υπάρχει Ευρώπη, διότι πάντα παρενέβαινε σε κρίσιμες ε, καταστάσεις, οπότε πάντα θεωρήθηκε ότι ήταν ένα θετικό μηχανισμός που όπως θα ήθελα να υπενθυμίσω παρεμβαίνει ώστε να προσφέρει αρρωγή στις προσπάθειες που κάνει ήδη το κράτος. Μιλάμε τώρα για χρονοδιαγράμματα και για ταχύτητα ενεργοποίησης. Η ταχύτητα ενεργοποίησης ε, σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η βοήθεια αυτή πολύ πιο γρήγορα. Εάν χρειάζεται πολύ χρόνο υπαρχει αυτών των κονδυλίων, ε, είναι λιγότερο ο χρόνο ε, εφαρμογή των σχετικών μηχανισμών αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο έτη χρόνο. Μέχρι να γίνει η αίτηση και μετά να δοθούν ε, τα κονδύλια στο κράτος μέλος και να είναι διαθέσιμα, περνάνε δύο χρόνια. Αυτό μας εμποδίζει στις ε, επεμβάσεις αποκατάστασης που χρειαζόμαστε νωρίτερα. Μειώνοντας λοιπόν τους χρόνους θα μειώσουμε το χρόνο που τελικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το, η βοήθεια αυτή. Κατά την άποψή μου το κράτος που υποβάλλει την αίτηση με ή χωρίς τα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέμβει, πρέπει να ανταποκριθεί ανεξάρτητα από το αν θα παρέμβει το Ταμείο Αλληλεγγύης. Το Ταμείο Λυγής, πιστεύουμε εμείς, ε, υποστηρίζει δαπάνες που ούτως ή άλλως το πληγέν κράτος πρέπει να ε, χρησιμοποιήσει διότι οι δραστηριότητες αρρωγής χρειάζονται άμεσα. Ένα μεγάλο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων μπορούν όπου υπάρχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας να κληρωθούν ε, αργότερα από το ε, ταμείο. Εμείς λοιπόν ε, δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα που τα κονδυλία διατίθεται 8-9 μήνες μετά από το αίτηση. Ο μηχανισμός συμμετοχής είναι σίγουρα χρήσιμος, αλλά πρέπει να δούμε ποιο είναι το πραγματικό ε, μέσο. Δεν είναι ότι εάν το Ταμείο Ελληνικής δεν παρέμβει δεν παρεμβαίνει και το κράτος. Το Ταμείο Ελληνικής υποστηρίζει το κράτος το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τις δραστηριότητες και το επιτρέπει να χρησιμοποιήσει και άλλους πόρους για την ανοικοδόμηση, για την αποκατάσταση. Όχι γιατί οι παρεμβάσεις είναι ανοικοδόμησης, διότι έχοντας πάρει την πρώτη βοήθεια το κράτος, μετά το ταμιολογής του προσφέρει προς τους πόρους για την, που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ανοικοδόμηση. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν τη σωστή διάσταση στο μηχανισμό αυτό με τις ε, απαραίτητες αναλύσεις. Ε, της κάθε αλλά βάσει των δικών μας εμπειριών αυτά είναι οι απόψεις μας για τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία θα υπάρξει ένας νέος κανονισμός ο οποίος θα αναθεωρήσει τα πράγματα. Να υπενθυμίσω τις φάσεις που προβλέπει ο τρέχον κανονισμός για την πρόσβαση στο Ταμείο και τη χρήση του. Να σας πω επ' αυτού κάποιες σκέψεις μας για κάθε φάση για το πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Όπως γνωρίζετε όλοι, ο κανονισμός προβλέπει μια φάση αίτησης. Οι φημισμένες 10 εβδομάδες από την αρχή του έτους, όπου το πληγέν κράτος συντάσσει το φάκελο αίτησης για πρόσβαση στο Ταμείο. Μετά υπάρχει η φάση αξιολόγηση από την Κομισιόν που απαιτεί περίπου 8-9 μήνες και μετά έχουμε την φάση υλοποίηση, το χρόνος αυτός κατά τον οποίο τα κονδυλία παρέχονται στο κράτος και το κράτος χρησιμοποιεί αυτά τα κονδύλια είτε για να, εμ, ως χρήματα επιστροφής ουσιαστικά που του παρέχονται για έξοδα που έχει ήδη κάτι ή για άλλες παρεμβάσεις, αποκατάστασης και μετά υπάρχει και μια φάση υποβολής έκθεσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι εδώ από αυτή την άποψη καλό είναι να δούμε τι θέλουμε, τι μορφή θέλουμε να έχει το μελλοντικό μέσο αυτό και κατά πόσο πρέπει να αλλάξουμε ορισμένα μέρη του. Σαφώ πρόσβαση στο Ταμείο έχουν τα κράτη-μέλη ε, και οι χώρε στο πλαίσιο βοήθεια. Ε, βοήθειας. Ε, σε περιπτώσει καταστροφών που αντιστοιχούν σε 3 δισεκατομμύρια σε σχέση με το ΑΕΠ. Υπάρχει λοιπόν κάποια συνοχή με τον νέο κανονισμό. Να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει με τον νέο κανονισμό. Όσον αφορά αυτό το major disaster, τη μείζωνα καταστροφή, υπάρχουν δύο εξαιρέσει. Η μία που επιτρέπει σε ε, χώρες γειτονικές με γειτονικά σύνορα που έχουν πληγεί από την ίδια καταστροφή να κάνουν αίτηση για κονδύλα και μετά η περιφερειακή υπόθεση, η δυνατότητα δηλαδή ότι αν δεν, φτάνει το, αν δεν επιτυγχάνεται το των τριών δισεκατομμύριων μια περιφέρεια που έχει πληγεί μπορεί να έχει πρόσβαση στο κονδύλια αυτά, παρότι η καταστροφή είναι μικρότερη, η ζημιά είναι μικρότερη από τα 3 δισεκατομμύρια. Και ήθελα να πω ότι εδώ αυτή τη στιγμή προβληματιζόμαστε κατά πόσο αυτά τα κριτήρια, τα ποσοτικά, ε, μήπως θα πρέπει να γίνουν ε, ποσοτικά. Στο σημερινό κανονισμό και αυτό έχει προβληματίσει πολλούς από όσους διαπραγματεύονται αυτόν τον νέο κανονισμό. Ε, ξεπερνάμε αυτή τη φάση κατά κάποιο τρόπο σήμερα για να υπερασπίσει κανεί περιφερει... Ε, μια καταστροφή σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχουν ε, επιπτώσει διαρκείας στην Ιταλία. Τις τρει αιτήσει πρόσβαση στο Ταμείο από το 2002 μέχρι σήμερα, οι 7 απορρίφθηκαν για σωστούς λόγους. Αυτές οι 7 που απορρίφθηκαν ήταν όλες περιφερειακής διάστασης διότι δεν αποδείχθηκε σαφώς ότι υπάρχει μακροχρόνια επίπτωση για την συγκεκριμένη περιφέρεια. Περνώντας λοιπόν από την ποιοτική προσέγγιση στην ποσοτική, είναι πολύ σημαντική μετάβαση για τις μελλοντικές ε, εφαρμογές του Ταμείου. Αφού ληφθεί λοιπόν τα κονδύλια, οι πόροι αυτοί πρέπει να κατευθυνθούν προς συγκεκριμένους τρόπους επεμβάσεων. Πέραν της αρρωγής προς τον πληγέντα πληθυσμό, για την οποία συμφωνούμε όλοι, προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεων αποκατάστασης των υποδομών που έχουν υποστεί ζημιά. Ήθελα λοιπόν εγώ να πω εδώ ότι αυτό δεν είναι ένα ταμείο πρόληψης, γιατί η πρόληψη καλό είναι να αφαιρώνεται σε άλλους, ε, ε, να βασίζεται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Από τα ταμεία συνοχής, ε, τα διαφορετικά ταμεία είναι πόροι που έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση από το Ταμείο Λιγκής. Το Ταμείο Λιγκής έχει διαδικασίες επιτρέψτε μου να πω, λιγότερο γραφειοκρατικές, ε, πιο ευέλικτες και γρήγορες, ενώ τα άλλα κονδύλια όπως το Ταμείο Συνοχής έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην πρόσβαση. Διότι η γραφειοκρατική διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη, ενώ το Ταμείο Αλληλεγγύης, παρότι εξακολουθεί να έχει κάποιους ε, περίπλοκους μηχανισμούς, ε, θεωρείται από όλους ένα πιο γρήγορο ταμείο, δηλαδή βρίσκεται πιο κοντά ε, στην ανταπόκριση. Ε, ε, Σαφώς κατά τη φάση εφαρμογής το ετών κράτος πρέπει να αποδείξει η υποδική του ευθύνη μια σειρά γεγονότων που αφορούν τις ζημίες βασισμένες σε συγκεκριμένα στοιχεία. Σήμερα με τον νέο κανονισμό γίνεται προσπάθεια να παρέχονται άλλου τύπου πληροφορίες, για παράδειγμα κατά πόσο υιοθετήθηκαν προληπτικά μέτρα στην πληγήσα περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται προσπάθεια να αποφύγουμε τον κίνδυνο της ε, της ε, μη παρέμβασης ουσιαστικά της προληπτικής παρέμβασης του κράτους σε αναμονή του Ταμείου Αλληλεγγύας αλλά πρέπει να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα δηλαδή όταν εγώ χρειάζεται να παρέμβω ε, για να διορθώσω κάτι, να αποκαταστήσω κάτι. Δεν μπορώ να πηγαίνω να ψάχνω να βρω κατά πόσο είχαν γίνει προληπτικέ δράσει προηγουμένω. Δεδομένη τη φύση τη καταστροφή, για παράδειγμα σε περίπτωση ενό σεισμού, όπω συνέβη στην Ιταλία, όπω συμβαίνει στην Ιταλία, όπου έχουμε ιστορικά κτίρια υπάρχει κίνδυνος ε, και επικινδυνότητα που για να προληφθεί χρειάζεται τεράστια κονδύλια. Εγώ λοιπόν στον επόμενο σεισμό δεν μπορώ να πω ότι θα έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα, διότι στον επόμενο σεισμό που θα γίνει στην Ιταλία υπάρχει κίνδυνος για θύματα και για σημαντικές ζημιές ε, σε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά μας που είναι εκτεθειμένη. Πώς να το κάνουμε. Ε, δηλαδή προληπτικά μέτρα είναι κάτι εξαιρετικά σύνθετο για μια τέτοια πολιτιστική κληρονομιά. Αν υπερχεί μια, ένας γεωλογικός κίνδυνος μπορεί να κάποια υποδομή να αντιμετωπιστεί. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, ε, μην επιβάλλουμε στα κράτη τα οποία υποβάλλουν κάποια αίτηση ε, να μας αποδείξουν πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να επαληθευτούν. Μετά έχουμε όλη τη διαδικασία πρόσβασης, αξιολόγησης ε, της Κομισιόν 8-9 μήνες όπως γνωρίζουμε. Σωστό είναι να υπάρχει μια τέτοια φάση αξιολόγησης. Και ο νέος κανονισμός θα μπορέσει να μας βοηθήσει εδώ. Θα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Κομισιόν και κράτους μέλους. Αυτό το διάστημα των 10 εβδομάδων από πολλούς θεωρείται σε μια γκυλοτίνα ουσιαστικά. Ε, εάν δεν προλάβει κανείς να τα κάνει όλα στις 10 εβδομάδες ε, βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Ε, αυτή λοιπόν την περίοδο ανταλλαγής, αξιολόγησης, σας την κάνουμε μια ε, περίοδο ανταλλαγής μεγάλης ε, πληροφοριών μεταξύ κρατούς μέλους και κομισιών. Ας ανοίξουμε λοιπόν την φάση αξιολόγησης και στο ενδεχόμενο του να γίνονται πολύ περισσότερες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ κρατούς μέλους και κομισιών που δεν πρόλαβαν να γίνουν στις πρώτες δέκα η φάση λοιπόν αξιολόγηση που θα μειωθεί ε, από του 8 μήνε στου 8 μήνε, α την ε, αξιολογήσουμε ώστε να εμπλουτίσουμε ένα φάκελο όποιο θα φαίνεται ε, ότι έχει λείψει στην αρχή. Και μετά υπάρχει και η φάση υλοποίηση. Αυτή τη στιγμή που λαμβάνουμε λοιπόν τα χρήματα, ξεκινούν οι δαπάνε. Και αυτή η φάση είναι σημαντική. Και μπορώ να σα πω ότι το έτος αυτό, αυτό το δεκάμινο, είναι ένα ικανοποιητικό διάστημα αλλά ίσως να μην αρκεί πάντα. Εγώ βέβαια μιλώ ως Ιταλός, εκ μέρους της Ιταλίας, ε, μια χώρα που για τους σεισμούς του Ισάκουλα χρησιμοποίησε 393 εκατομμύρια, για την Εμίλια Ρωμάνια πάνω από 650 εκατομμύρια. Όταν αξοδεύκανε σε 650 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο, ε, θα φτάσω στο συμπέρασμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σύνθετο θέμα. Προσοχή λοιπόν με τα χρονοδιαγράμματα γιατί είναι πολύ σύνθετο το θέμα. Και μετά υπάρχει και ο γνωστός μηχανισμός ε, σύμβασης που ε, θέλουμε να μειώσουμε. Υπάρχει ένα άλλο σημαντικό έγγραφο που είναι το Annual Report, της έκθεση που βασίζεται σε πληροφορίες των κρατών μελών ε, ε, αυτό το annual report λοιπόν ε, θα βοηθήσει και στη διαμόρφωση του νέου κανονισμού και ελπίζω και στο μέλλον ε, θα πράξει το ίδιο. Όπω θα δείτε η Ιταλία χρησιμοποίησε σχεδόν τη μισή χρηματοδότηση που έχει παρασχεθεί. Αυτά είναι τα σημαντικότερα γεγονότα, τα πιο πρόσφατα θα έλεγα. Είτε αναφερόμαστε σε major disaster είτε σε regional disaster όπου η Ιταλία έλαβε χρηματοδότηση αυτό που αναπτύξαμε εμείς για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο Ταμείο και εδώ ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε Ήθελα να πω ότι αυτή μας εμπειρία από το 2002 επέτρεψε να οριμάσει στη χώρα μας επίσης ε, και αυτή η συνείδηση, η ευαισθητοποίηση που σχετίζεται με μια ομοιόμορφη μέθοδο αναγνώρισης της ζημίας ε, που πριν κάποια χρόνια δεν ήταν τόσο άμεση ε, δεν ήταν βασισμένη σε τόσο σαφείς κανόνες με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι για την αποκατάσταση της κατάστασης και από αυτούς μπορούμε να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ζημιές που έχουν λάβει χώρα, τους όρους από τους οποίους ε, έχει γίνει η αξιολόγηση του εκαστού κινδύνου κτλ. Αυτό μας επέτρεψε λοιπόν να εμβαθύνουμε και να, κάνουμε, να βελτιώσουμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση. Ευχαριστώ. Ε, thanks a lot, ε, Mr. D'Angelo. Σας ευχαριστούμε κύριε D'Angelo. Τώρα, δώσω το λόγο στην κυρία Φεραγκού, την εισηγήτρια. Το πρωί έγινε η ψηφοφορία για την έκθεσή σας. Αν μπορέσετε κύριε Φεραγκούτη να μας εξηγήσετε επομένω τα βασικά σημεία της εκθέσεώς σας. Και στη συνέχεια θα έχουμε τις ε, ερωτήσεις προς τους ε, εμπειρογνώμονες και κατόπιν δώσουμε το λόγο στους και και βουλευτές. Έχετε το λόγο να μας εξηγήσετε. Πρώτα πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ειδικού και εμπειρογνώμονες για όλες αυτές τις πληροφορίες στην ακρόαση. Σήμερα το πρωί σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε το κείμενο. Η αναθεώρηση του Ταμείου Λεγγύης Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετική μεταρρύθμιση και οπότε ακούσαμε την Επιτροπή των Περιφερειών, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε διάφορες ε, συμβαστικές τροπολογίες, περίπου 60 γενικά τροπολογίες υποβλήθηκαν και όπως είπαν και οι ειδικοί πήγαμε τις 15 εβδομάδες όσον αφορά τις ε, αιτήσει και επίσης ε, από 12 σε 18 μήνες το διάστημα της ε, υλοποίησης. Ε, είπαμε επίσης και για την ε, τεχνική αρρωγή που προσφέρει το Ταμείο, επίσης και για τις προκαταβολές. Έχουμε τώρα αξιοποιεί από κάποιους νομικούς φραγμούς για τις πλήγησες χώρες. Επίσης είπαμε για 1% του ΕΠ θα οριστεί το Ταμείο είχε πει 1,5% η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς έχουμε 1% και έτσι τώρα να καλύπτεται καλύτερα ένα τέτοιο φαινόμενο μιας θεομηνίας και επίσης νομίζω απλουστεύσαμε σημαντικά τη διαδικασία ούτως ώστε να διορθώσουμε κάποια δύνατα σημεία που είχαν εμφανιστεί όλα αυτά τα χρόνια που ισχύει ο εν λόγω κανονισμός. Βέβαια, τα κακά μαντάτα είναι ότι έγιναν περικοπέ από τον προπολογισμό όσον αφορά την προϋποδότηση του Ταμείου. Άρα, τώρα θα έχουμε λιγότερα χρήματα. Πάντω θα πρέπει να συνεχίσουμε κάθε Και έτσι θα γίνει ο πρώτο τρίλογο στι 12 Φεβρουαρίου, 19 και 24 επόμενε συναντήσει. Οπότε θα πρέπει για να συμφωνήσουμε όλοι να επιδείξουν ε, κάποια ευελιξία και να πάει στο Μάρτιο στην Ολομέλεια η έκθεση ήδη. Έχουμε κανονίσει τις συναντήσεις με την Ελληνική Προεδρία. Σήμερα το πρωί ήρθε εδώ ο Έλληνας υπουργό και μας είπε ότι πρόκειται για μία από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας, το Ταμείο Αλληλεγγύης. Επίσης, υπάρχει ένα για το 1,5% και το 1%. Κάποιοι στο Συμβούλιο θεωρούν ότι ε, κάποιες ότι θα, θα πρέπει να δοθεί 1,5% από τις χώρες, άλλοι λένε 1% θα βγει κάτι από τις ε, ε, Πάντως έχουμε πλημμύρες, έχουμε ξηρασίε, έχουμε δηλαδή κάποιες καταστροφές που κρατούν αρκετό χρόνο. Γι' αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει να παραταθούν οι σχετικές ε, προθεσμίες. Πάντως θα πρέπει να δοθεί κάποια ευελιξία στην όλη διαδικασία. Επίσης, Yo creo que el Parlamento ha hecho un buen trabajo y... Είπαμε ότι από την ονοματολογία και οι χώρες ε, του ΝΑΤ 3 και του ΝΑΤ 2 μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Όλοι πάντως εδώ ήταν χρήσιμο που σας ακούσαμε γιατί διευκρινίστηκαν πολλά πράγματα. Και κάτσε και σημείωσε ένα σωρό πράγματα και είμαι σίγουρη ότι όλα όσα άκουσα σήμερα από εσά θα είναι πολύ χρήσιμα για τι διαπραγματεύσει. Thanks a lot. If you have... Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χρυσόγελο. Τώρα, εάν έχετε κάποιε ερωτήσει, τρει ή τέσσερι, ε, και κατόπιν έχουμε σύντομε απαντήσει από του ειδικού, και κατόπιν να ε, γίνει συζήτηση, να προλάβουν το λόγο και οι ισχυρότερε ηγητές και οι άλλοι βουλευτέ. Πώ αν θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Okay. okay, so are there some questions? Έχετε ερωτήσεις. Έχετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ναι, έχω κάποιες ε, παρατηρήσεις και κατόπιν μια ερώτηση. Βεβαίω και ήταν πάρα πολύ θετικό το έργο τη Ρώσα με έκθεσή τη. Νομίζουμε το θέμα ήταν επίγοντο χαρακτήρα. Επίση, Εγώ ως Γαλλίδα έζησα την καταστροφή που υπέστη η Βρετανία αλλά και η Ιρλανδία και η Μεγάλη Βρετανία και στο βάρ της Νοτιού Γαλλίας επίσης είχαμε βροχή κατρακτώδη πάνω από 20 ώρες οπότε είχαμε αγνοωμένους έναν ε, νεκρό ε, πάνω από χίλιους α, οι οποίοι έπρεπε να διασωθούν. Οπότε μπορούμε να θυμηθούμε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλές θεομηνίες και βέβαια ακόμα δυστυχώς οικοδομούμε στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Άρα πρέπει να γίνεται διάγνωση κάθε φορά του εδάφους. Χρειάζεται μέσα αυτό το πολιτέ πρόγραμμα των μιζώνων κινδύνων. Αυτό το, έτσι το ονομάζουμε στην Γαλλία, έχει μορφή νόμου και αυτό έχει να κάνει επίσης με τις ε, αναγκαστικού χαρακτήρα εγκρίσεις για οικοδόμηση. Βεβαίω η Ευρώπη εδώ μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο. Φυσικά και η Επιτροπή μας επίσης αρμοδιότητα, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια του Ταμείου ελληνική για να βοηθήσει αυτούς που έχουν πληγεί. Βεβαίω και σωστό να γίνει απλούστευση διαδικασία, διαδικασίας. Στόχοι είναι να έχουμε ευελιξία, να έχουμε αποτελεσματικότητα και επίσης έχουν γίνει κάποιες προτάσεις μεταρρυθμίσεων του κανονισμού για να πετύχουν αυτούς στόχους και κατά τη γνώμη μου πρώτος σημαντικός στόχος και σημαντικός είναι να έχουμε μια γενική συμφωνία σε θελουσία βάση για να έχουμε καλύτερο συντονισμό και παρέμβαση. Να παρέχετε βοήθεια αμέσως μας χτυπήσει η καταστροφή. Και είπαμε ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ανταλλαγή πληροφοριών ούτως ώστε να μην γίνονται τα ίδια λάθη από όλα τα κράτη. Αλλά και τα περιφερειακά ταμεία θα πρέπει να βοηθήσουν και στην προληπτική αντιμετώπιση. Να έχουμε κάποια έργα υποδομής, να έχουμε κάποια διασυνοριακά κονδύλια. Βλέπουμε ότι έχουμε όλο περισσότερες θεομηνίες. Χρειάζεται επομένω περισσότερη συνεργασία. Πυροσβέστες, ε, διασώστες, νοσοκομιακά, ό,τι χρειάζεται. Είπαμε για συνειδητοποίηση. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε επομένω. Ό,τι μπορούμε και αυτή η μεταρρύθμιση του οργανισμού να βοηθήσει στην Ολομέλεια του Ιανουαρίου είχα υποβάλει μια προφορική ερώτηση στις 6 Φεβρουαρίου έχουμε παρέμβαση της επιτροπές Νομίζω ότι όλα τα ερωτήματα τα οποία αναδύονται από το κείμενο της Ρώσα απαιτούν άμεση απάντηση. ε... Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Αν θέλετε να τοποθετηθείτε, να αντιδράσετε σε κάτι που ακούσατε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάποια σχόλια ή κάποιες τοποθετήσεις από πλευράς μου. Για συγκεκριμένες συστάσεις ε, <clears throat> της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αναφέρεται η σπουδαιότητα της κοινωνίας των πολιτών, οι εθελοντικές δράσεις και δομές που είναι πολύ σημαντικές μετά την καταστροφή θεομηνία. Προτείνουμε συμπεριληφθεί αυτού του είδους η πολιτική πρωτοβουλία ανάληψη δράσης ε, από την κοινωνία των πολιτών στο σύστημα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης και των Δράσεων. Πρώτο σχόλιο αυτό. Δεύτερον, θα είχα κάποια ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω προς την κυρία Φεραγκούτ συγκεκριμένες συστάσεις ε, που επικεντρώνονται στην αναδάσωση μετά από πυρκαγιές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της αναδάσωσης για τα δάση και βραχυπρόθεσμα να αρχίσει άμεσα η αναδάσωση που είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα για τις νότιες περιοχές της Γαλλίας, Προβάνση, το νότο της Ευρώπης γενικά στις χώρες του νότου και είναι λοιπόν σημαντικό να αναφερθεί αυτό το θέμα της αναδάσωσης. Έχω αυτό το ερώτημα. Θα συμφωνούσατε λοιπόν για αυτή την ε, περιβαλλοντική σπουδαιότητα της αναδάσωσης που πρέπει να συμπεριλαμβάνεται. Ευχαριστώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πράγματι, το θέμα αυτό προσπαθήσαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων για τις τροπολογίες γινόταν ε, λόγος ε, στην αρχή της έκθεσης για ξηρασία, για πλημμύρες, για πυρκαγιές στο τέλος όμως της διαπραγματεύσεις αυτό που θελήσαμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα γενικό εδάφιο για καταστροφές θεομηνίες μακράς διάρκειας, χωρίς να εξειδικεύσουμε τη μία την άλλη. Υπήρχαν πολλές τροπολογίες για κάθε μία από τις θεομηνίες ή καταστροφές. Υπήρξε λοιπόν αυτή η γενική αναφορά η κάλυψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε περίπτωση πυρκαγιών η δυνατότητα να αποκατασταθεί το αρχικό τοπίο με αναδάσωση συνεπάγεται εμπλοκή της αναδάσωσης ως δράσης. Και αυτό σε σχέση με αναδασωση συνεπαγεται εμπλοκη τη αναδασωσης ως δραση και αυτο σε σχεση με με τις του Ταμείου Αλληλεγγύης. Λαμβάνω υπόψη και δέχομαι αυτή την πρόταση, διότι είναι απαραίτητο το θέμα της αναδάσωσης στις περιπτώσεις πυρκαγιών και το θέμα της εθελοντικής υπηρεσίας για την κοινωνία των πολιτών εθελοντικού χαρακτήρα ε, συνεισφορά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Ευχαριστώ. Any other Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν, παρατηρήσεις. Ωραία, λοιπόν. Κάποια σχόλια μόνο. Ήμουν εγώ εισηγητή εξ ονόματος των Πρασίνων και θα ήθελα κάπως να υπεξηγήσω κάποια θετικά στοιχεία ε, σε σχέση με την έκθεση αυτή. Θα μιλήσω ελληνικά τώρα, ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι μετά από 7 χρόνια στην πραγματικότητα που είχε μπλοκάρει η διαδικασία είμαστε τώρα ε, πολύ πιο κοντά στο να υιοθετηθεί η, η, νέα, η νέα ρύθμιση για το Ταμείο είναι σημαντικό γιατί όπως αναφέρθηκε και πιο πριν το Ταμείο αυτό αναδεικνύει την Ευρώπη της αλληλεγγύης δηλαδή ότι η Ευρώπη είναι παρούσα όταν συμβαίνει μια καταστροφή αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί βάζει και τη διάσταση της ανάγκης να πάρουμε προληπτικά μέτρα για να μην πληρώνουμε συνέχεια καταστροφές δηλαδή ότι υπάρχει αυτή η διάσταση ότι Πρέπει να μαθαίνουμε από τα παθήματά μας για να μην ερχόμαστε συνέχεια να πληρώνουμε καταστροφές. Είτε αυτό αφορά τις πλημμύρες ή άλλες ε, περιστάσεις, γιατί πολλές φορές είναι τα ίδια λάθη που οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Ε, είναι σημαντικό επίσης ότι αναγνωρίζουμε ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα εξαιτία κλιματικής αλλαγής και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την κλιματική αλλαγή αλλά και την ανάγκη προσαρμογής στα νέα δεδομένα είτε αυτό αφορούν, ε, τα θέματα των πλημμυρών ή τα θέματα των καταστροφών, πυρκαγιών κλπ. Είναι σημαντικό να επανασχεδιάσουμε στη βάση της πρόληψης του κινδύνου, ε, όπως αναφέρθηκε και από την ε, κυρία Σάντσες Σμιτ, για παράδειγμα πρέπει να ξέρουμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες, ποιες έχουν χτιστεί πάνω σε περιοχές που κινδυνεύουν και οι κίνδυνοι σήμερα έχουν μεγιστοποιηθεί. Δηλαδή είχαμε μια, ένα λάθος σχεδιασμό. Κατασκευάσαμε πολλές φορές κοντά σε ποτάμια, κοντά σε ε, επικίνδυνες περιοχές κτίρια και σήμερα αυτός ο κίνδυνος μεγαλώνει εξαιτία κλιματικής αλλαγής. Άρα έχουμε δύο παράγοντες που επιδεινώνουν το πρόβλημα και θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο νομίζω είναι σημαντικό είναι η προσέγγιση του οικοσυστήματος, τα θέματα αποκατάστασης. Δηλαδή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν είναι μόνο θέμα τεχνικής, δεν είναι μόνο θέμα πολιτικών μηχανικών, αλλά μιας νέας αντίληψης ε, που λαμβάνει υπόψη την προσέγγιση του οικοστήματος για να κάνουμε σωστά έργα αποκατάστασης. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, επίσης, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι αποσαφηνίζονται οι κανόνες. Πολλές περιφέρειες και πολλά κράτη είχαν μια ε, θολή εικόνα για το ποια, προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Τώρα είναι πολύ πιο σαφείς οι κανόνες. Ε, είναι ε, ενδιαφέρον ότι επιταχύνονται και οι διαδικασίες απάντησης αν είναι επιλέξιμο ή όχι ε, ένα έργο αποκατάστασης από το Ταμείο αυτό το διάστημα του ενός μήνα που πρέπει να απαντηθεί η οχι ενα εργο αποκαταστασης απο ενός κράτους μέλους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην υπάρχει μια σύγχυση γύρω από το αν είναι ή όχι επιλέξιμο, ότι ορίστηκαν ε, διαδικασίες επιτάχυνσης αλλά μέσα σε λογικά χρονικά όρια για όλες τις διαδικασίες και αποκατάστασης και πληρωμής από το Ταμείο. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή έκθεση και δεν είναι τυχαίο ότι πήρε πολύ μεγάλη υποστήριξη σχεδόν ομόφωνη από την Επιτροπή ε, πολύ μικρή ήταν η αποστασιοποίηση. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε τώρα με το Συμβούλιο και με την ε, Κομισιόν μέσα από τον τρίλογο στις τρεις αυτές συναντήσεις, ώστε πράγματι να επιταχυνθεί μέσα στο Φεβρουάριο η διαδικασία και να υπάρχει μια συμφωνία γιατί και οι πολίτες και οι περιφέρειες και η κοινωνία των πολιτών περιμένουν ένα αποτέλεσμα πάνω σε αυτή την έκθεση και σε πάνω σε αυτό το ταμείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν ε, σχόλια, θα ήθελα να τοποθετηθεί η Κομισιόν. Θέλετε να απαντήσετε σε κάτι. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και αυτήν εδώ την Επιτροπή και τους εμπειρογνώμονες ε, η εμπειρία των οποίων κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση της Κομισιόν. Όσον αφορά τη διαχείριση αυτού του μηχανισμού τα τελευταία σχεδόν 12 χρόνια. Αληθεύει ότι το Ταμείο μέχρι στιγμής ε, έχει παρουσιάσει κάποιες αδυναμίες. Αυτές έχουν εν μέρει να κάνουν ε, με την ταχύτητα με την οποία χρειάστηκε να δημιουργηθεί το 2002 ως άμεση ε, ανταπόκριση ουσιαστικά σε ένα επίγον περιστατικό της εποχής. Όπως θα θυμάστε, η Κομισιόν προσπάθησε να βελτιώσει το μηχανισμό αυτό ήδη από τα πρώτα χρόνια. Ίσως να υπήρξε υπερβολικά φιλόδοξη εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία 2005 δεν ήταν επιτυχής. Αυτή τη φορά λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε το υπάρχον ταμείο παραμένοντας εντός του συστήματος, δηλαδή να κάνουμε κάποιες προσαρμογές στον υπάρχοντα κανονισμό χωρίς να προσθέτουμε εντελώς νέα στοιχεία στον κανονισμό αυτό και κυρίως χωρίς ε, να προσθέτουμε επιπλέον δυνατότητες δαπανών. Αντιθέτως το ταμείο μειώνεται από ένα δις σε 500 εκατομμύρια ετησίως. Ε, σε αυτό το πλαίσιο θα χρειαστεί να ε, δράσουμε. Και η προσέγγιση που αναφέρεται αφορά ενδεχομένω μια πλήρη αλλαγή του συστήματος. Ε, ίσως όμως να μην είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν πρέπει να υπεφορτώνουμε το ταμείο που υπάρχει σήμερα με άλλες πολιτικές όπως πρόληψη κτλ. Είναι απολύτως σαφές ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική και το ταμείο πρέπει να θεωρείτε ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλειών της Κομισιόν. Το Ταμείο Λεγγύης από μόνο του δεν δύναται να χειριστεί τα πάντα. Υπάρχουν τα διαρθρωτικά ταμεία όπου αποτελούν προτεραιότητα οι προληπτικές πολιτικές. Υπάρχουν ε, πρωτοβουλίες ε, στο περιβαλλοντικό ε, τομέα, υπάρχουν πρωτοβουλίες πρόληψης από την Κομισιόν. Εάν δείτε λοιπόν το Ταμείο σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι το Ταμείο όντως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά στο συγκεκριμένο τομέα για τον οποίο έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιεί οικονομικά τα κράτη-μέλη. Να βοηθά οικονομικά, συγγνώμη, τα κράτη-μέλη ανταποκρινόμενο σε καταστροφές. Ανεξάρτητα των διαδικασιών πρόληψης και τα λοιπά. Ο κύριος Γιάξης ανέφερε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είπατε θα ήταν σημαντικό τα κρατημέλη να γνωρίζουν ε, σε πολύ πρώιμο στάδιο κατά πόσο το Ταμείο θα μπορέσει να επισέλθει, να ενεργοποιηθεί και κατά πόσο οι δικαιούχοι μπορούν να υπολογίζουν σε οικονομική στήριξη. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση που έχουμε μπροστά μα αυτή τη στιγμή για τον κανονισμό θα οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Εμεί προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε εφόσον υιοθετηθεί έτσι, ε, προσπαθήσαμε να ορίσουμε πιο σαφή κριτήρια που θα επιτρέπουν σε ένα κράτο μέλο ευθύ εξ αρχή να γνωρίζει κατά πόσο υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να λάβει τέτοια χρηματοδότηση. Διότι σαφώ εάν ε, δεν πληρούνται τα κριτήρια θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να λάβει. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να είναι απόλυτα σαφή στο μέλλον. Και ειδικότερα εφόσον έχει γίνει μια προκαταβολή όπως αυτή που προτείνουμε η πιθανότητα επέμβασης του Ταμείου ε, αυξάνεται ουσιαστικά με ασφάλεια 100% σχεδόν μπορεί να πιστεύει το κράτος μόλις θα λάβει τα κονδύλια αυτά. αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thanks a lot. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνουμε ένα 15 λεπτό διάλειμμα και στις 4.30 θα υποδεχθούμε εδώ σε αυτή την αίθουσα τον Επιτρόπο, τον κύριο Γιώχανες Χάν, για να συζητήσουμε μαζί του την τρέχουσα κατάσταση της ε, πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, I think we, we, we can't wait anymore for the rest of the... δεν περιμένουμε για να έρθουν και οι υπόλοιποι, οπότε να μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε αυτό το ε, σημείο και παρακαλώ όλοι όσοι θέλετε να μιλήσετε, να αποχωρήσετε. Έχουμε τώρα τον Επίτροπο τον κύριο Γιώχανε Χάν, ο οποίο θα μα μιλήσει, θα ε, μα εξηγήσει πού βρισκόμαστε όσον αφορά ε, την συγκρότηση τη νέα ε, πολιτική συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, ευθύς αμέσως κύριε Επιτροπή, μπορείτε να μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα. Μήπως ε, για την κάμερα είναι καλύτερα το διπλάνο. δεν πειράζει, αν το, έχω το ετοιμάσετε το μικρόφωνο. Δεν πειράζει, έτσι θα έχουμε το ίδιο μικρόφωνο. Καλό είναι αυτό. Δείχνει ότι είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για, την... για το ότι με προσκαλέσατε πάλι να παραστώ ενώπιον σας και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το όπως έχουν εξελιχθεί οι συζητήσεις και οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ώστε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ενημέρωση και για τα operational programs, τα λειτουργικά προγράμματα. Και υπό αυτό το πρίσμα και πνεύμα να αναφερθώ στις προπαρασκευές. Είχατε σήμερα την δυνατότητα να συζητήσετε τα θέματα των κατεξουσιοδότηση πράξεων, delegated acts. Θα ήθελα να σας κάνω λόγο για την ρήτρα επενδύσεων και για το πώς έχει σήμερα η παγκόσμια συνιστόση, η παγκόσμια διάσταση για αυτό το θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτική μας εκτός Ευρώπης και αυτό είναι κάτι που από κοινού εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτό το γεγονός. Είναι επιτυχία στην ενημέρωση, στην επικοινωνία και πληροφόρηση και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, Ήδη το 2012, πάνω από ένα χρόνο ήδη παλαιότερα, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να γίνει ένας άτυπος διάλογος για την χρήση των κονδυλίων για τα κονδύλια των διαθωτικών ταμείων και την χρήση κονδυλίων ώστε να μην χάσουμε χρόνο μετά την ας το πω έτσι επίσημη έναρξη ε, των δράσεων το 2014 και μπορώ να πω ότι έγιναν δεκτές αυτές οι προτάσεις ε, για έναν άτυπο διάλογο και το αποτέλεσμα σήμερα είναι τρεις επίσημες τρεις επίσημες partnership agreements, συμφωνίες εταιρικής σχέσης που βρίσκονται ήδη στο ε, θεσμικό μας όργανο. Τρεις. Και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες τον μεγάλο αριθμό των ε, συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, θα τον έχουμε στα χέρια μας, τις πρόσθετες προτάσεις και σε ένα αυξημένο, προηγμένο επίπεδο. Και αυτό στο τέλος τέλος θα δίνει την δυνατότητα ταχύτερης εφαρμογής και υλοποίησης και κυρίως ε, αυτών των συμφωνιών από πλευράς μας. Αναμένουμε από πλευράς της Επιτροπής όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτές τις διατάξεις εταιρική σχέσης και να τις καταθέσουν κατά την Άνοιξη. Και σύντομα αμέσως μετά να περάσουμε στα λειτουργικά προγράμματα και αμέσως ε, σε παράλληλη ε, διαδρομή να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Λογικά εξαρτώνται βέβαια τα πράγματα από τα κράτη-μέλη. Όταν τα πράγματα θα έχουν οριμάσει και θα έχουν υποβληθεί προγράμματα και σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνει ένας έλεγχος ποιότητας ώστε να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρίνονται στις διατάξεις και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, αυτά τα σχέδια. Οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις είναι η επικέντρωση των κονδυλίων σε στοχοθετημένους στόχους και προηγούμενες εκ προημίου εξάντε προϋποθέσεις και διατάξεις που πρέπει να υλοποιούνται. Και σε διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη ακριβώς αυτές οι διατάξεις και αυτό το πλαίσιο αυτών των εταιρικών σχέσεων θα μπορέσουν να διαμορφώσουν προγράμματα λειτουργικά που θα αρχίσουν να λειτουργούν. Δεν αποκρύπτω ότι στοχεύουμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, κατά τη, αυτές τις συμφωνίες κατά τη διάρκεια της δικής μας εντολής ε, να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε. Και απλά και μόνο για να καταφέρουμε γιατί διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος στη μεταβατική περίοδο να καταλήξουν και να υπάρξουν λόγω καθυστερήσεων, λόγω της αλλαγής ε, ε, ε, του πλαισίου και της Επιτροπής να υπάρξουν καθυστερήσεις. Ενώ πρέπει να γίνουν γοργά τα πράγματα. Αυτό όμως εξαρτάται από τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και από την προπαρασκευή και προετοιμασία όσον αφορά τα έγγραφα για το σχεδιασμό και είναι σημαντικό και θέλω και πάλι να το τονίσω αυτό, ότι η ποιότητα, η ποιότητα έχει πρωτεύοντα ρόλο εναντί της ταχύτητας. Πρώτα η ποιότητα, μετά η ταχύτητα δεν θέλουμε να υπάρξει πίεση αν ε, στο τέλος πρέπει άμεσα γοργά να αποφασιστεί κάτι βιαστικά. Όχι. Η ποιότητα έχει πρωτεύοντα ρόλο έναντι της ταχύτητας. Διότι μιλάμε για ένα χρονορίζοντα δεκαετών ετών de facto εκ των πραγμάτων. Και τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεκαετών, ετών, δεκαετή περίοδο, ένας μήνας παραπάνω ή παρακάτω δεν μπορεί να είναι αποφασιστική σημασία για την ποιότητα του προ, ενός προγράμματος ή σχεδίου για τις, κατη, για τις κατεξουσιοδότηση ε, πράξεις που αποτελούν αντικείμενο εξέτασης από την Ευρωβουλή καταρχήν θα ήθελα να πω και δεν μπορούμε να το κάνουμε αρκετά συχνά ότι σε σχέση με την ε, έγκριση του πλαισίου για την πολιτική συνοχή θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Ήταν μια μακρά διαδικασία αλλά στέφθηκε με επιτυχία στο τέλος τέλος και για την πολιτική συνοχή είναι ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα αυτό. Πρέπει να διασφαλίσουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία και στιγμή όχι μόνο τα αναγκαία μέσα και εργαλεία να είναι στη διάθεσή μας αλλά αυτή η πολιτική να μπορέσει μέσα σε νέα πλαίσια μέσα σε νέες δομές να υλοποιηθεί. Η συζήτηση για τις κατεξουσιοδότηση πράξης και κατεντολήν πράξης έχουν το, ξεκίνησαν το 2013 από το πλαίσιο συζητήσεων των ομάδων επαϊόντων και ειδικών μέσα στο πλαίσιο της, ε, ε, των εντολών για τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Τότε ξεκίνησαν αυτές οι διαβουλεύσεις. Υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα στοιχεία όλων των συνεδριάσεων ώστε να είναι ενήμερο το Ευρωκοινοβούλιο Κοινοβούλιο για το τι συμβαίνει πάντα σε σχέση με αυτέ τι διαβουλεύσεις. Για τις συζητήσεις για τις εξουσιοδότηση πράξη, κατά εξουσιοδότηση πράξης, προσκαλείται το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετέχει στι συνεδριάσει των επαϊόντων, των πραγματογνωμόνων και από ό,τι γνωρίζω έχει συμμετάσχει ήδη η Ευρωβουλή σε πολλές από αυτές τις ε, διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις. Είναι προς το συμφέρον όλων το νομικό πλαίσιο γοργότερα, το δυνατόν γοργότερα να ολοκληρωθεί, ώστε οι σημαντικότερες κατεξουσιοδότηση πράξεις να διαβιβάζονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διαβιβαστούν πριν από την περίοδο ευρωεκλογών, ώστε να μπορέσουμε σε αυτό το πεδίο να κάνουμε πολλά πράγματα όσον αφορά την περίοδο που απομένει στη διάθεσή μας και να διευθετήσουμε, να διεκπαιρεώσουμε πολλές υποθέσεις. Σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι εξουσιοδοτήσεις για το συνολικό πακέτο το, της πολιτικής συνοχής να ε, κατανεμηθούν σε πέντε πράξεις ε, ώστε να μπορέσουν να δημοσιευθούν έγκαιρα και με τις εξής προτεραιότητες. Πρώτη προτεραιότητα Πρώτη προτεραιότητα για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις ε, για έναν Ευρωπαϊκό Δεοντολογικό Κώδικα για τις εταιρικές σχέσεις. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκριθεί αυτό σήμερα, από ό,τι ακούω, υπάρχει μια διεξοδική και πολύ θετική συζήτηση, σε βάθος συζήτηση, για αυτό το σχέδιο από πλευράς της Επιτροπής μας. Θέλω να τονίσω λοιπόν εδώ ότι εκφράζω την ικανοποίησή μου και ευελπιστώ ότι αυτές οι νομικές πράξεις που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το πλαίσιο, ότι γνωρίζουμε ότι για το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι ένα πολύ σημαντικό ε, έγγραφο αυτό. Αυτή τη στιγμή κατεξουσιοδότηση εξουσιοδότηση πράξης συμπεριλαμβάνουν διαφορετικά θέματα για τον προγραμματισμό, το αποθεματικό επιδόσεων, την, διακυβέρνηση, ε, την μορφή ε, διαχείρισης ε, και την δυνατότητα μετακύλησης. Η εξουσιοδότηση και όσον αφορά τον κανονισμό αποτελεί τμήμα αυτού του πακέτου δράσεων. Στοχεύουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη δεύτερη δέσμη κατ' εδώ πράξεων κατά τα μέσα Φεβρουαρίου να ε, την καταθέσουμε. Και αν τα καταφέρουμε πριν από την ε, εκπνοή της εντολής του Ευρωκοινοβουλίου, πριν από τις ευρωεκλογές, θα θέλαμε το Ευρωκοινοβούλιο να πάρει την τρίτη δέσμη, το τέταρτο, την τέταρτη δέσμη που ε, εμπεριέχει λιγότερο κατεπήγοντα θέματα, θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο στη συνέχεια. Αυτές οι πράξεις σας περιλαμβάνουν τις εξουσιοδοτήσεις για ιδιωτικές και δημόσιες συμπράξεις ώστε να αποφευθούν ατυπίες, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αριθμίες και προβλήματα. Αυτές οι κατεξουσιοδότηση πράξεις που ιστερότερα θα κατατεθούν θα καλύπτουν τις εξή πτυχές. Την εισαγωγή κατά ποσών για κάποιους τομείς. Ε, δείκτες ε, όσον αφορά τις εκθέσεις ε, που θα συντάσσονται και κατά αποκοπήν πάλι ποσά τα οποία θα συσχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συνοψίζω, γνωρίζουμε όλοι ότι αν δεν καταφέρουμε να τα καλύψουμε αυτά και να ασχίσουν να ισχύουν πριν από την εκπνοή της εντολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του 2014 με τις ανάλογες επιπτώσεις που θα συνεπάγονται αυτές οι καθυστερήσεις. Γι' αυτό καταβάλει αναγκαίες προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να προετοιμαστούν αυτά τα έγγραφα έγκαιρα. Τώρα, δύο λόγια για το θέμα της ρήτρα επενδύσεων, της επενδυτικής ρήτρα. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι το ύψος των επενδύσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται σε ένα ενδεδειγμένο επαρκές ύψος. Οι επενδύσεις μέσα στο πλαίσιο των διαθωτικών ταμείων πρέπει να λειτουργούν ώστε να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη οι δημόσιες επενδύσεις θα έχουν ρόλο κλειδιού σε αυτό το πλαίσιο σε σχέση και με τις ιδιωτικές τίνουν ε, να αυξήσουν ε, τα μερίσματα και την κερδοφορία των κεφαλαίων. Σε μια περίοδο ύφεση ε, οι δημόσιες επενδύσεις υποστηρίζουν ιδιαίτερα και μπορούν να συνδράμουν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ένα ειδικό πλαίσιο. Με αυτή τη συγκυρία της κρίσης οι δημόσιες επενδύσεις βλέπουμε ότι συρρυκνώνονται, μειώνονται στην Ευρώπη και δυστυχώς έχουν φτάσει σε ένα χαμηλό επίπεδο ρεκόρ σε ένα ναδύρ ε, και γι' αυτό τα προγράμματα της ε, πολιτικής συνοχής λόγω της, του περιορισμού των δημοσίων δαπανών και λόγω του, των διατάξεων της, του Συμφώνου ε, Ανάπτυξης ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε προληπτικά να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο για την, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα κράτη-μέλη, για τον υπολογισμό των προσπαθειών που πρέπει να γίνουν ώστε να καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να μειωθούν κιόλα. Και έτσι η ένταση μεταξύ δημόσιων ελλημάτων θα μειωθεί και θα υπάρξει δυνατότητα ανάκαμψης και ανάπτυξης ε, με τις ε, δαπάνες αυτές που θα διασφαλιστούν. Αυτή η προσέγγιση νομίζω είναι συνετή και λογική. Δύο λόγια παραπέρα ακόμα για τη διεθνή διάσταση της πολιτικής συνοχής αυτή η διεθνής διάσταση της πολιτικής συνοχής κατά τα τελευταία έτη ενισχύθηκε σημαντικά. Είναι μια επιπρόσθετη ευκαιρία αυτή να έχουμε νέες καινοτόμε μορφές συνεργασίας, συνεργασίας με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα αλληλοδιάδοχα σχέδια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των προπαρασκευαστικών δράσεων ε, μπορούν να ενισχυθούν με αυτά τα κονδύλια και αυτές τις δράσεις. Ευχαριστώ την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, για την υποστήριξη που μας έχει δώσει. Σήμερα ο διάλογος για την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική των πόλεων αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση με 10 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα με χώρες στρατηγικούς εταίρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Βραζιλία, Κίνα, Ρωσία ή και η Ιαπωνία μεταξύ αυτών. Στα ισχυρότερα επιχειρήματά μας αυτές οι συζητήσεις ποια είναι. Είναι η διεθνής πολιτική πείρα που έχουμε συλλέξει ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε υπέρ των περιφερειών αμφωτέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Να μπορέσουμε το πλαίσιο ενίσχυσης και υποστήριξης και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την ενδυναμώσουμε και την αξιοπιστία στον ιδιωτικό τομέα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβουλές για παράδειγμα που μπορούν να χορηγηθούν, τεχνογνωσία ουσία εξαγωγή ε, αυτών των ε, στοιχείων και στην περίπτωση της περιφερειακής ανάπτυξης να συναχθούν συμπεράσματα με βάση Πόσο ο ανταγωνισμός για παράδειγμα και οι ε, εντολές και οι ε, συμβάσεις θα μπορούν να ε, συνεισφέρουν υπέρ των συντελεστών της αηφόρου ανάπτυξης και της πρόθεσης και της δημοκρατίας. Στη Βραζιλία το πρότυπο της βραζιλιάνικης περιφερικής ανάπτυξης έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα όσον αφορά τους στόχους και τα συστήματα υποστήριξης πλαίσια ώστε έχουμε και πολλά σεμινάρια που έχουν γίνει για τέτοια προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγής, προγράμματα αποστολών που έχουν διοργανωθεί σε σχέση με τη Βραζιλία. Το ίδιο ισχύει ακριβώς και για τον τομέα της ε, ισχυρής ε, έντονης ανάπτυξης, ε, όπου ιδιαίτερα η Κίνα, η Ιαπωνία, αλλά και κάποιες χώρες της Λατινικής, της Νότιας Αμερικής, για λόγους που μπορεί κανείς να υποθέσει και μπορεί να ε, γνωρίζει τις προσδοκίες σε σχέση με αυτούς ε, μπορούν να προωθηθούν. Λάβαμε υπόψη με ικανοποίηση ότι η Περιφερειακή Επιτροπή έχει ε, εγκρίνει την ε, έκθεση, το, η ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο συνεχίζει τις εργασίες για το σχέδιο ε, από πλευράς μας και ελπίζουμε ότι αυτή η επικαιροποίηση θα μπορέσει ε, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές να εγκριθεί. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που από το 2005 το παρακολουθούμε και ασχολούμεθα με αυτό. Διαρκώς αναφύεται όταν έχουμε προβλήματα θεομηνιών και καταστροφών για το Ευρωπαϊκό Αναφέρομαι Ταμείο Αλληλεγγύη και θα πρέπει εδώ να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε ευρύτατες διαβουλεύσεις ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ε, τύχει ευρείας ε, έγκρισης ε, αυτή το το σχέδιο και πρέπει να είναι δυνατόν με επιταχυμένους γοργότερους ρυθμούς να παρέχουμε τη συνδρομή μας ε, σε όσους πλήττονται από τέτοια φαινόμενα και να υπάρχει και καλύτερη εκτίμηση από πλευράς των κρατών μελών αν ε, κάτι είναι επιλέξιμο ως σχέδιο και μπορεί να υποστηριχθεί ή όχι και πρέπει να συνεισφέρουμε για να μπορούμε άμεσα ταχύτερα να αντιδρούμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Να ρωτήσω πρώτα τους συντονιστές, ε, δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Ωραία λοιπόν εσείς πρώτα και μετά η Κωνσταντσε. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση για όλους μας ε, πιστεύω. Να υποβάλω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη που αφορά το σημείο κλειδί της, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης. Οι πληροφορίες είναι σαφείς για να είμαι ειλικρινής διότι κάποιες χώρες και οι άλλες στο μέλλον υπάρχει και πιο έγγραφο θα υπάρξει κάποιο έγγραφο σύντομα το έχουμε ήδη συζητήσει ένα έγγραφο στο οποίο να μπορούμε να διαβάσουμε για αυτή την πρόοδο και περισσότερο για το περιεχόμενο γιατί οι μεγάλες αλλαγές ε, είναι η αιρεσιμότητα εξάντε, νέα χρηματοδοτικά μέσα, συνέργειες ε, Έχουμε τα στρατηγικά έγγραφα. Θα ήθελα εγώ να γνωρίζω περισσότερα γιατί είναι πολύ καλά τα νέα που μας φέρατε σήμερα. Δεν πειράζει αν αργήσουν τα πράγματα αυτά για μερικούς μήνες, αλλά μετά εσείς έχετε φύγει. Θέλω λοιπόν να ακούσω λίγο τη δέσμευσή σας. Μια ερώτηση κάνω, μην γελάτε να σας πω ότι η Επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου ήδη προτίθεται να οργανώσει μια ακρόαση σε ένα-δυο μήνες από τώρα για να ακούσει τις απόψεις των διαφορών εταίρων. Όπως είπατε, συμφωνήσαμε για αυτή την κατεξοδότηση πράξη για τον κώδικα διοντολογίας και η ερώτηση είναι έχει υλοποιηθεί είναι ουσιαστικά αυτή μια νέα διαδικασία σχεδιασμού και συνεργασίας όχι μόνο εντός της χώρας αλλά ενίοτε και για την εξέβρεση των σωστών εταίρων μέσω της έξιμης εξειδίκευσης εκτός της χώρας. Πώς προχωράνε αυτές οι διαδικασίες. Καλό θα ήταν να έχουμε την ευκαιρία να δούμε και πιο λεπτομερώς τις επιδόσεις. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το γεγονός ότι Έχουμε λιγότερα χρήματα από ό,τι αναμέναμε. Έχουμε μεγάλα προβλήματα μπροστά μας ε, όσον αφορά τις ε, ικανότητες πληρωμών ε, που θα έχουμε στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής μπορείτε να μας ενημερώσετε γι' αυτό δεν υπάρχει πρόβλημα υπάρχουν πολλά λεφτά που θα δούμε του χρόνου Γιατί αν έρθουν θα λύσουμε το πρόβλημα πληρωμής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των νέων, ε, της ανεργίας. Υπάρχουν λοιπόν στόχοι να πιέσετε περισσότερο τα κράτη-μέλη εκείνα που ήταν επιφυλακτικά. Και μετά είπαστε ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι με τη συγχρηματοδότηση. Εκπληκτικό. Ωστόσο, ορίσαμε συγκεκριμένα ποσοστά στους κανονισμούς. Τι εννοείται λοιπόν ευέλιξία προς τα κάτω ή προς το πάνω. Πώς το εννοείτε. Και μετά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα διότι το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί, το δημόσιο σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα, αλλά αν δώσετε διασφαλίσεις για κάποια έργα, ίσως ε, άλλοι χρηματοδότες όπως οι τράπεζες να αναλάβουν την ευθύνη όπως έκαναν πριν από την κρίση. Και γι' αυτό θα, θα, θα με ενδιαφέρει να ακούσω κάτι, ποια πράγματα περισσότερα. Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την σωστή επικοινωνία. Διότι εδώ τα πράγματα δεν βρίσκονται σε φυσιολογική ροή όπως τη γνωρίζαμε. Έχουν αλλάξει μέθοδοι, έχουν αλλάξει στόχοι, έχουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μήπως μαζί με τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να οργανώσουμε μια εκστρατεία το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο Καταλαβαίνετε γιατί ζητάω. Για να γίνουν τα πράγματα πιο γνωστά στους πολίτες, ότι αυτή είναι η πολιτική με τις μεγαλύτερες επενδύσεις για περιφέρειες, για πόλεις, για αγροτικές περιοχές. είμαστε, έχουμε παραμείνει σιωπηροί ε, άνθρωποι. Και φυσικά ε, καταλαβαίνω, ξέρετε ακολουθώ και τα tweet σας στο Twitter, αλλά είναι πολύ καλά. Αλλά τι γίνεται με όλα αυτά τα μεγάλα έργα που θα μπορούσαμε να δημοσιοποιήσουμε ώστε να πούνε οι άνθρωποι ναι θα σας ψηφίσουμε. Αυτά γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δεν πάω να θεωρώ ότι έχετε κάνει εκπληκτικό έργο. Μα υποστηρίξατε σε όλε τι διαπραγματεύσει. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με την τρέχουσα κατάσταση. Απλά λόγω των φιλοδοξιών που είχαμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το θέμα όσο το περισσότερο εντό αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, Κωνσταντζ. Η κυρία Κράιλ, ευχαριστώ πολύ Ντανούτα. Κάποιες ερωτήσεις θα είχα και εγώ. Θα με ενδιέφερε πράγματι να δούμε ποιες είναι αυτές οι τρεις χώρες που πάνε μπροστά ως πρωτοπόρες. Είπε ο Γιάννη ότι η Πολωνία είναι μία από αυτές. Θα ήθελα, το ξέρω αυτό για την περίπτωση αυτή, θα ήθελα να μάθω για τις άλλες δύο. Κυρίως για το θέμα του αν συμπεριλαμβάνεται ένα από τα κράτη-μέλη που έχει ένα ιδιαίτερο υψηλά, υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων. Και θα έθετα το ερώτημα, υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες απόψεις πώς για τους νέους, την απασχόληση για τους νέους Youth Employment Initiative μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Ήταν αίτημα του Κοινοβουλίου το δυνατόν ταχύτερα να λειτουργήσουν τέτοια σχέδια και προγράμματα. Αλλά πρέπει να εξαρτάται και από τις ε, συμφωνίες εταιρική ε, σχέσεις ε, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό. Με ενδιαφέρει να ξέρω, κάναμε αυτό το βήμα προς τα εμπρός. Δεύτερο, όταν έχουμε τέτοιες συμφωνίες εταιρικής σχέσης και αναμένουμε τις επόμενες σε μικρό χρονικό διάστημα σύντομα προσεχώς, αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη αυτών των συμφωνιών βαίνει εκ παραλίλου με την έγκριση των κανονισμών από πλευράς μας. Με ενδιαφέρει να μάθω με ποια βάση αυτές οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν κατατιστεί και έχουν γίνει. Με βάση την παλαιότερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τουλάχιστον έχουν ενταχθεί στο νέο πνεύμα των κανονισμών και διατάξεων που τον ε, Δεκέμβριο τελικά εγκρίναμε εμείς ε, καθοριστικά. Μπορεί κανείς να πει σε σχέση με τον δεοντολογικό κώδικα ότι εντάξει υπήρξαν δεσμεύσεις στις διαπραγματεύσεις ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα αντανακλούν αυτό το πνεύμα. Εντάξει, ωραία Α το πω έτσι, από πλευρά των προτάσεων των κρατών μελών για τέτοια σχέδια θα μπορείτε να αξιολογήσετε αν πραγματικά συμβαίνει αυτό ή όχι ή αν πιθανώς ίσως θα πρέπει να υπάρξουν να καλυφθούν με περαιτέρω έργο το οποίο θα πρέπει να γίνει από πλευρά μα, να καλυφθούν αυτέ οι ανάγκε. Και κάτι τελευταίο, ίσω μπορεί να αναγνωρίσει κανεί ότι υπάρχει ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη που έχουν κάποιε σημαντικότερε δυσκολίε εφέτο να καταλήξουν σε τέτοιε συμφωνίε εταιρική σχέση. Είτε επειδή δεν έχουν την επαρκώ τη δύναμη, την ικανότητα να ε, εφαρμόσουν τη νέα πολιτική συνοχή ε, στη χώρα του, ε, στρατηγικέ προσεγγίσει που θα πρέπει έπρεπε να εφαρμοστούν είτε επειδή φαίνεται ότι ίσως τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να μπορούν να κάνουν ταχύτερα τις ε, δράσεις τους και τις, ε, τα καθήκοντά τους για να μπορούν να υποβάλουν τέτοιες προτάσεις και τέτοια σχέδια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τον λόγο και εγώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είχα δύο ερωτήσεις και μάλιστα ξεκινώ λέγοντας με την πρώτη ερώτηση κατά την έγκριση των κανονισμών έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό που έχει εγκριθεί. Δηλαδή η ελαστικότητα που πρέπει να διασφαλίζεται σε σχέση με την μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των κυριότερων προτεραιοτήτων ή αξώνων. Θα με ενδιέφερε να γνωρίζω κατά πόσον αυτό είναι κάτι που αποτελεί αντικείμενο που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη ως μέσο. Δεύτερη ερώτηση. Οι νέες διατάξεις από πλευράς κανονιστικού πλαισίου θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ένα μέρος των κονδυλίων θα χρησιμοποιείται για την καινοτομία, την έρευνα, την ανάπτυξη. Έτσι δεν είναι. Και πρέπει να χρησιμοποιούνται για αυτούς τους στόχους, για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Και επίσης να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται και για μια επιρροή που πρέπει να μπορεί να ασκείται με τις ε, περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές και περιφέρειες αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια προς αυτή την κατεύθυνση. Με ενδιαφέρει να μάθω γίνεται αυτό ή όχι. Thank you and για τους πράσινους. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ από πλευράς μου να τονίσω και να πω πως οι δύο εισηγητές να γνωρίζω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά μεριμνά και διασφαλίζει ότι τα πράγματα αυτά θα λειτουργούν με το επίκαιρο, επικαιροποιημένο πλαίσιο του κανονισμού. Από όσα είδα εγώ σε σχέση με σχέδια που έχουν κατατεθεί δεν συμβαίνει αυτό, αλλά το έγγραφο του Συμβουλίου, η θέση του Συμβουλίου είναι το θεμέλιο για αυτή τη δουλειά, για αυτό το έργο. Υπάρχουν μικρές ε, διαφορές και διαφοροποιήσεις όμως και θα θέλαμε αυτές ε, οι διαφοροποιήσεις να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις θέσεις του Συμβουλίου. Παράλληλα με τον δεοντολογικό κώδικα θέλω να αναφέρω στο ότι πρέπει να είναι σαφές το πώς θα λειτουργεί η διαδικασία σε λεπτομέρειες σε σχέση με το άρθρο 14 σαφέστατες επισημάνσεις ε, για το τι πρέπει να εμπεριέχεται σε αυτό το πλαίσιο και δεύτερον, επίσης καταφέραμε τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να δημοσιοποιείται προηγούμενα ε, σε σχέση με την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν μπορούν όλα αυτά να διασφαλιστούν και αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά και να ε, πιστοποιηθούν ότι οι αναγκαίες διαδικασίες ε, στα αντίστοιχα άρθρα στο 7 και στο 8 δηλαδή θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες όπως προβλέπετε ιδιαίτερα όσον αφορά το tracking. Και θέλω να το επισημάνω και να πω ότι εδώ υπάρχει μια κατεξουσιοδότηση πράξη που ήθελε να εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει ακόμα αυτή. Και υποθέτουμε ότι σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να υπάρξει μια νέα επεξεργασία και μάλιστα με ιδιαίτερο ζήλο για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Συγκεκριμένα θα ήθελα να μου πείτε, αληθεύει αυτό το οποίο ακούμε από εσά επίτροπε, ότι η δική σας διοικητική αρχή, δηλαδή για τα περιφερειακά θέματα, στις διαβουλεύσεις των κρατών μελών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επικαιροποιημένη έκδοση του κανονισμού, ώστε να προετοιμάζονται τα αντίστοιχα έγγραφα. Διότι με εκπλήσει ότι κράτη-μέλη καταθέτουν σχέδια και έγγραφα και ε, έντυπα όπου ενώ έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο για τον κανονισμό, για τις κανονιστικές διατάξεις δεν λαμβάνονται αυτές πλήρως υπόψη. Αυτές αντανακλώνται όπως θα έπρεπε ναι ή όχι. Δεύτερο που με ενδιαφέρει είναι αυτό το οποίο είπατε για τη ρήτρα επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη θέση της πρέπει να πω ότι δεν κατανοώ απόλυτα ποια θα είναι η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως θα ακολουθηθεί τώρα. Θα μπορούσατε να τη διευκρινίσετε σας παρακαλώ. Uh, thank you, Commissioner. Ευχαριστούμε. Επίτροπε, έχετε τώρα το λόγο. Μάλιστα. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τις συμφωνητερικές σχέσεις θα πρέπει να σας πω ότι το 2012 τελευταίο τρίμηνο δώσαμε αυτό το έγγραφο τοποθέτηση, όπως το λέμε στα κρατή-μέλη, και έτσι ήταν προσβάσιμη σε όλους η, κατάσταση για όλες τις υπηρεσίες τη επιτροπή τι γίνεται όσον αφορά τη χρήση των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό φορούσε κάθε κράτο μέλο και επί τη βάση αυτών των εγγράφων έγιναν οι διαπραγματεύσει. Οπότε και κατά τις διαπραγματεύσεις ανεφίεσαν και άλλα ζητήματα, συζητήσεις, σχέδια κειμένου και όλα αυτά προετοίμασαν, προδίκασαν αν θέλετε την κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Τις επόμενες εβδομάδες ε, και το μήνα των επόμενων θέλετε Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι στοιχείο, ό,τι πληροφορίες θέλετε. Δεν γίνεται όμως να δημοσιεύσω, να, να, να διαβιβάσω όλα τα email τα οποία συνόδευσαν ε, αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και τα κρατημέλη επίσης έχουν δημοσιοποιήσει ε, τις θέσεις τους για τις ε, διαπραγματεύσεις. Α, Φερρυπίν έχω κατά τώρα την Πολωνία, οπότε και έτσι θα δείτε τι γίνεται. Έχουμε, είπαμε, τρεις χώρες οι οποίε ε, ε, τα έχουν δημοσιεύσει ήδη, ξέρουμε, Λετωνία και Γαλλία είναι οι άλλες δύο και Λιθουανία, Φιλανδία, Σλοβακία, Σουηδία ε, αναμένονται τις αμέσως επόμενες μέρες και όσον αφορά τις ε, πληρωμές, μάλιστα, δεν πρέπει να δώσω και ο Γενικός Διευθυντής σήμερα είπε τα επικαιροποιημένα στοιχεία, είπε ότι πρόκειται για 60 δις από πέρυσι. Οι 16, 16, 16, πρόκειται για κάποιες αξιώσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί μετά το τέλος Οκτωβρίου. Άρα είμαστε μέσα στην προθεσμία των 60 ημερών. Όμως θα υπάρξει πρόβλημα περί τα τέλη του έτους γιατί γίνεται έτσι μια σόρευση, μαζεύονται Ξέρετε την κατάσταση, τα κράτη-μέλη ουδέποτε απεδέχθησαν την πρότασή μας για συμπληρωματικό προϋπολογισμό. για αυτές τις συγκεκριμένες αξιώσεις πληρωμών. Οπότε δεύτερο ίμιση του έτους προκύπτουν κάποια προβλήματα. Όμως Εμεί ελπίζουμε ότι θα εξυπηρετήσουμε τι αξιώσει κατά του πρώτου μήνε του 2013, λέει ο Επίτροπο. Τώρα, όσον αφορά την ερήτρα επενδύσεων, πρόκειται για ένα εργαλείο, για μια ευκαιρία για τα κράτη-μέλη, εκείνα τα οποία δεν βρίσκονται στην διαδικασία του υπερβάλλοντος ελλείμματος, οπότε είναι δυνατόν να γίνει κάποιο είδους ε, αφαίρεση της εθνικής συγχρηματοδότησης από το έλλειμμα. Διότι νομίζω ότι έχουμε κοινό συμφέρον να γίνουν επενδύσεις και είναι κάπως γελίο να μην μπορεί να γίνει κάποια επένδυση λόγω του κινδύνου να ξεπεραστεί το όριο του ελλείμματος. Οπότε και οι χώρες εκείνες που δεν έχουν ε, περιβάλλον έλλειμμα, είπαμε, όλες οι υπηρεσίες να του δώσουν την ευκαιρία να κάνουμε μια τέτοια είδους ε, αφαίρεση της ε, εθνικής συγχρηματοδότησης από το έλλειμμα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να συμφωνείτε και μια χρονιά μετά την άλλη κάθε χρόνο. Υποβάλλεται έτοιμα και γίνεται κατά περίπτωση η δικασία να δοθεί η έγκριση όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα το οποίο υποβλήθηκε μια ερώτηση όντως σε κάποια κρατημέλη ακόμα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την πρόσβαση στην δανειοδότηση. και τα συναφή. Οπότε δεν είναι τώρα το πρόβλημα μόνο προδοσιμότητος, αλλά είναι και η τεράστια διαφορά που υπάρχει στα επιτόκια από τη μία χώρα στην άλλη. Και πολλές φορές αυτό γίνεται σε χώρες που είναι πάρα πολύ κοντά. Ας πούμε, μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας. Τα εταιρικά δάνεια, όσον αφορά το επιτόκιο, είναι 4-5% στην Ιταλία και στην Ελλάδα ακόμα είναι 7-8% για τα εταιρικά δάνεια. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε συγκροτήσει μια ομάδα εργασία για το ζήτημα τούτο. Διότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον όπου τα διευθυντικά ταμεία θα χρησιμοποιηθούν περισσότερο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του μετοχικού κεφαλαίου. Γιατί πάρα πολλέ χώρε δεν μπορούν να πάρουν γιατί δεν μπορούν να ε, παράσχουν εγγύσει υπό τον τύπο του μετοχικού κεφαλαίου, ε, περιουσιακά στοιχεία εταιρεία κλπ. Οπότε, σύντομα προτείνω να διεκδοθούν κάποιε προτάσει, διότι σε κάποιες χώρες ακόμα υπάρχουν ευκαιρίες κανείς να ε, πάει τα λεφτά του. Βέβαια έχουμε κάποια ταμεία για τις ΜΜΕ και ότι ακόμα υπάρχει ευκαιρία, υπάρχουν κάποια, κάποια χρήματα για τους ε, επιλέξιμους. Οπότε έτσι μπορούμε να έχουμε κάποιες ευκαιρίες επενδυτικές. Έχετε δίκιο για την επικοινωνία. Αυτό είναι αιώνιο. Ε, κυρίως θέλω να δω τι θα γίνει με κάποιες χώρες όπου τα διαρκικά ταμεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και να δούμε τι γίνεται επιτόπου στο κάθε κράτος, να δούμε τι, τι λένε οι αρμόδιοι υπουργοί, να τους παρουσιάσουμε μια, ένα σύμφωνο εταιρική σχέση, να δούμε τι πιθανότητες υπάρχουν και επίσης για ε, άλλοι συνάδελφοι που δεν είναι μέλη της Περιφερικής Επιτροπής σας θα πρέπει να διαδώσουν αυτή μας την πολιτική στις χώρες τους. Είναι σημαντική η πολιτική αυτή και θα πρέπει να επενθυμίζουμε, θα πρέπει να τονίζουμε ότι έχουμε αλλάξει την κατεύθυνση της πολιτικής, δεν την εστιάζουμε στις ε, υποδομές, αλλά ε, την εστιάζουμε τώρα στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και τα τα ταμεία έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά το κρατικό τομέα, ούτως ώστε να δώσουν λύσεις για την κρίση, για την έλλειψη χρημάτων. Και έτσι μπορεί να διπλασιαστούν τα χρήματα τα οποία υπάρχουν για την ε, στήριξη της οικονομίας από τα 70 δις 2007-2013 και πάμε στα 240 δις για τις προοπτικές 2014-2020 και βεβαίως θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση μετά τις περικοπές που είχαν στον προϋπολογισμό, στους προϋπολογισμούς. Ό,τι γίνεται, ό,τι είναι δυνατόν να γίνει. για τις πρωτοβουλίες για την απασχόληση των νέων. Αυτή τη στιγμή λίγα πράγματα μπορώ να σας αναφέρω, γιατί βρίσκεται στις αρμοδιότητες της απασχόλησης, ε, του τομέα απασχόλησης. Ε, και εδώ σε σχέση με την εφαρμογή των ε, πραγμάτων δεν μπορώ να αναφέρω κάτι. Καταρχήν θέλω να επαναλάβω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις για τις ε, συμφωνίες για τις εταιρικές ε, σχέσεις φυσικά χαρακτηρίζονται με ιδιαίτερο τρόπο από την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και στόχος ήταν της χρήσης των κονδυλίων έτσι να γίνουν οι διαπραγματεύσεις υπό αυτό το πρίσμα Τώρα, να δει κανεί ε, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων στο Κοινοβούλιο και την ε, εφαρμογή τους ε, σε πρακτική μορφή και να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει η δυνατότητα υλοποίησης, θα έχουμε μια αξιολόγηση που θα κάνουμε. Αξιολόγηση με προθεσμία τέλη 2015 νομίζω, με διορία αλλά έχει ζητηθεί στον τομέα του δεοντολογικού κώδικα να συνταχθεί έκθεση για το τι, τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει και θέλουμε να διατηρήσουμε την πολιτική πίεση πολιτική πίεση. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε και δίνω συνέχεια σε αυτό. Σε κάποια κράτη φυσικά είναι διαφορετική η υλοποίηση και πρέπει να εντατοποιηθεί. Αυτό συσχετίζεται με την κατάσταση σε κάποια κράτη-μέλη όπου υπάρχει υψηλότερος βαθμός αποκέντρωσης αποκεντροποίησης και περισσότεροι εμπλεκόμενοι μπορούν να εντάσσονται έτσι σε αυτό το πλαίσιο. Ενώ σε άλλα κράτη που έχουν κεντροποιημένες δομές έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Εμπλέκονται περισσότερο οργανώσεις, σύλλογοι και δομές που βρίσκονται άμεσα κάτω από το κεντρικό διοικητικό ε, διαχειριστικό επίπεδο στο κράτος και έχουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά, να καλυφθούν οι περισσότεροι. Παρακολουθούμε τα πράγματα, θα συνταχθεί έκθεση στο τέλος και θα ασκηθεί πίεση πολιτικά ώστε να προαχθεί αυτό το θέμα όπως, όπως μπορεί να γίνει. Και σε σχέση με τις εταιρικές ε, συμφωνίες, εταιρικής σχέσης, για μια χώρα όπου μπορεί να έχει κάποιες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζει είναι κατανοητό όμως αυτό. Είναι η Κροατία αυτή η χώρα όπου εδώ ε, είναι ιδιαίτερα απασχολημένοι με ιδιαίτερα έντονο τρόπο να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ένταξης, πώς να το πω, τις, τα προγράμματα και φάσεις ε, στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτά. Μην το ξεχνάμε, μέχρι τα, μέχρι τα μέσα του 2013 ήταν προενταξιακή χώρα. Μετά για ένα εξάμεινο ήταν πλήρες μέλος. Και τώρα έχουμε τη νέα περίοδο που ξεκινά και πρέπει να παρακολουθήσουν και να συμμορφωθούν σε αυτήν. Έχουν προβλήματα δυναμικού και προσαρμογής δυναμικού. Και διτά, διότι υπάρχει, είναι μια χώρα που έχει, είναι αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων για όσα τεκταίνονται εκεί. Μπορούμε να κατανοήσουμε όμως ότι συμβαίνουν και σημειώνονται κάποιες καθυστερήσεις εκεί και υποστηρίζουμε και ε, ε, βοηθούμε τους Κροάτες να ξεπεράσουν αυτές τις στενοπούς και αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα τώρα σε σχέση με την ελαστικότητα χρησιμοποιείται αυτό το 10% κύριε Ευρωβουλευτά ώστε να έχουμε τη νέα κατεύθυνση τα κονδύλια στις πρωτεύουσες των περιφερειών να ε, εμβάζονται όσον αφορά και τη χρήση για την έρευνα. Γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το πλαίσιο, αυτή η δυνατότητα. Μια και τα νεότερα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν τα προβλήματα που υφίστανται. Ότι δηλαδή έχουμε περιφέρειες που ε, μπορούν να θεωρηθούν more developed regions και είναι κατανοητό ότι υπάρχει και συμπίκνωση εκεί επικέντρωση ερευνητικών δραστηριοτήτων όπως πανεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων. Εδώ και hardware και software και λογισμικό δηλαδή ε, για παράδειγμα πρέπει να μπορεί να εντάσσεται ώστε να ε, εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της ρήτρας ελαστικότητας και να χρησιμοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Προσπάθησα <clears throat> σε σχέση με τη ρήτρα επενδύσεων να αναφέρω τα σχετικά. Τώρα αν τα κατάφερα και είναι αρκετά σαφή τα πράγματα, μέχρι σήμερα η Ιταλία και η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία, αν τα θυμάμαι καλά και μπορώ από μνήμης να τα συνοψίσω περιληπτικά, έκαναν χρήση αυτής της δυνατότητας ή θα κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας υποβάλλοντας αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε οι εθνικές δαπάνες να μπορούν να συνυπολογίζονται μέσα στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης και να αφαιρούνται από το έλλειμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρία Θα Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μια πολύ απλή και ίσως όμως και δύσκολη ερώτηση θα ήθελα να διατυπώσω. Στον κανονισμό αυτό υπάρχει η επιλογή θεματολογικά να ενταχθεί η σφαιρική ε, ευρυζωνική προσέγγιση. Παρακαλούμε η ευρωζωνική αυτή επέκταση πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει στις χώρες μας. Όχι μόνο στα αστικά κέντρα αλλά και στο χώρο της υπαίθρου να μπορεί να προσφερθεί. Γι' αυτό η ερώτησή μου δεν θα σας εκπλήξει. Συχνά την αναφέρουμε στις εταιρικές συμφωνίες εταιρικέ σχέσης που θα συνταχθούν, θα καταρτιστούν, θα πρέπει να προβλέπετε και θα προβλέπετε ότι για τη Γερμανία, για παράδειγμα, θα πρέπει να ισχύει η ευρυζωνική υποστήριξη ε, ότι δεν θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ε, ενταχθεί. Φυσικά όμως έχουμε τη Γερμανία, στη Γερμανία πολυμορφία περιφερειών και πολυσχηδείς, πολύμορφες ε, δομές και διαρθρώσεις και έχουμε, για παράδειγμα, θα ήταν αρνητικό αν δεν θα μπορούσαν να υποστηριχθούν αυτές οι περιφέρειες, διότι η επέκταση του ευρυζωνικού φάσματος δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο πόλεις αλλά αφορά και περιφέρειες και ε, γι' αυτό η παράκλησή μου είναι, αν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ώστε σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις θα προβλέπετε ότι η ευρυζωνική υποστήριξη δεν θα συμπεριλαμβάνεται για τη Γερμανία από πλευράς του κανονισμού, γιατί τα ομοσπονδα κρατήρια, τα ομοσπονδιακά κρατήρια δεν μπορούν τα ίδια να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιούνται από, από το ένα μέσο ή από το άλλο και να επιλέγουν τα ομοσπονδιακά κρατήρια το τι θα γίνεται. Θα ήταν μια εφικτή διαδικασία αυτή, θα μπορούσε να λειτουργήσει λειτουργήσει για τη Γερμανία. Η αρμόδια, οι εμπλεκόμενοι ε, που είναι στο επίπεδο αυτό θα ήταν οι άμεσα αρμόδιοι θα μπορούσαν να επιλέγουν. Ευχαριστώ. Uh, thank you. Ευχαριστούμε. Μαρίτερε Σάντσε Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επανέρχομαι στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Ζητώ συγγνώμη κύριε Επιτρόπε, αλλά είναι τρει συμφωνίε που αποτελούν το αντικείμενο επίσημων προτάσεων είναι λίγο. Μπήκαμε στην νέα δημοσιονομική περίοδο, έχουμε νέα προγράμματα το 2014, γιατί μόνο τρει. Τι έχει καθυστερήσει, υπάρχουν προσκόμματα στις περισσότερες συμφωνίες εταιρικής σχέσης ή οφείλεται αυτό σε καθυστερήσεις των κριτικών μηχανισμών γιατί γνωρίζω ότι οι συμφωνίες είχαν ξεκινήσει να μελετώνται πριν από πολλούς μήνες. Ξέρω ότι στη Γαλλία η Κομισιόν έκανε παρατηρήσεις στη γαλλική κυβέρνηση. Την επέπληξε λόγω λοιπού σκέψης και στρατηγικής σε αυτές τις συμφωνίες τερικές σχέσεις και υπάρχει μια νέα πρόταση. Ανισχώ λοιπόν όσον αφορά την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων το 2014 θα είναι ένα κενό έτος όσον αφορά την υλοποίηση των έργων εφόσον δεν έχουν οριστεί τα επιχειρησιακά σχέδια και οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, τα έργα δεν μπορούν να υποβληθούν ε, στις περιφερειές ε, δεν θα χορηγηθούν κονδύλια εσείς έχετε υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα των επενδύσεων και των ταμείων την αγκαιότητα, το πόσο σπανίζουν τα δημόσια κονδύλια. Είναι πολύ αναμενόμενο αυτά τα κονδύλια στις περιφέρειες. Κάτι δεύτερο, ήθελα να επιθυμίσω ότι όλο και περισσότερο, κυρίως στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στα κράτη, ε, προωθείται ο πολιτισμός, αποτελεί σημαντικό κομμάτι του του χώρου προϊόντος αφορά τους νέους ε, έχουμε μελετήσει για διάφορα πολιτιστικά σχέδια εσείς ε, γνωρίζετε κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί αυτό το θέμα σε επιχειρησιακά προγράμματα και διασυνοριακά έχω την ίδια ερώτηση γνωρίζετε καθόλου κατά πόσο λαμβάνει προτεραιότητα αυτό το θέμα σε ορισμένες διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης ευχαριστώ, ευχαριστώ Μαριτερές Γιάννη Μπρέχτ Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια σειρά ομιλιών. Πρώτα πρώτα. Γύρω Ντέφα, που ήταν πολύ ενδιαφέροντα ομιλία μα πει, αλλά επίση ακούσαμε και τι γίνεται όσον αφορά αυτό το, το, το, το έλλειμμα, αυτό το κενό στι πληρωμέ για το 2013 όσον αφορά την πολιτική συνοχή, που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι το θέμα τι θα γίνει με τι ε, πληρωμέ, αν θα ικανοποιηθούν οι σχετικέ αξιώσει. Οπότε το ερώτημα είναι τώρα. Έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα του τοπίου. Γιατί οι πληροφορίε που έχουμε από τον Επιτρόπο Λεβαντόφσκι έφτασε σε εμά μέσω τη ε, επιτροπή προπολογισμών για αυτά τα 18 δι, νομίζω είναι λίγο τρομακτικό το πώ. Ε, πριν δε τη μεσημερινή διακοπή ήρθε ο Υπουργό ο κ. Χατζηδάκη και μα είπε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει μια δέσμευση μέτρων σε σχέση με τις ε, κατεξοδότητες πράξεις και το πρόβλημα είναι ότι κάποιες χώρες μέλη δεν είναι έτοιμες ε, να δεχθούν, δεν προτίθεται να δεχθούν κάποιες αυτές τις πράξεις. Ίσως μας είπε ότι θα γίνουν τρεις-τέσσερις από αυτές. Μας είπε τι πρόκειται για, για τρεις πράξεις, πρόκειται για ένα πακέτο. Γιατί, συγγνώμη, σου, είπε ο κύριο ε, Χαζηδάκη, η ελληνική προεδρία έχει πρόβλημα με αυτό το θέμα. Για πέστε μα εσεί πώ έχει η κατάσταση. Ευχαριστώ, Γιάννη. Ο Ιωάχιμ Τσέλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τα όσα μας εκθέσατε. Εγώ σχεδόν τίνω, πρέπει να πω, Δηλαδή, θετικό σημείο και πρόσημο να βλέπω στο ότι μόνο τρεις χώρες αυτές τις, ε, τα σχέδια για τις εταιρικές σχέσεις τα έχουν καταθέσει. Τότε θα υπήρχε η ελπίδα, λέω εγώ, ότι θα είχαμε πρώτα τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου και τις συμφωνίες με το Συμβούλιο που θα καταρτιστούν και θα συναυθούν και μετά θα είναι βάσεις αυτές οι συμφωνίες για τέτοιου είδους εταιρικέ σχέσεις. Και έτσι θα δημιουργηθούν τα λειτουργικά προγράμματα που θα λειτουργήσουν και φυσικά αυτό ισχύει και για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις που αναμένονται από πλευράς της Επιτροπής, ώστε να υπάρξει περαιτέρω αποσαφήνιση για την εφαρμογή όλων αυτών. Αυτή είναι η θετική ελπίδα που έχω, η αισιοδοξία μου. Από την άλλη πλευρά όλο και περισσότερα μηνύματα παίρνω ότι εδώ και μήνες εδώ με ζήλο και επιμέλεια εργάζονται επιτόπου οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με βάση τα σχέδια της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκλειστικά συζητούν και διαβουλεύονται με τους αρμόδιους επιτόπου όσον αφορά την κατάρτιση λειτουργικών προγραμμάτων. Είχαμε όμως συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ότι το δυνατόν περισσότεροι φορείς για τέτοιου είδους σχέδια, ιδιαίτερα από το τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να εμπλέκονται σε αυτές τις διαβουλεύσεις για να δίνουν τις απόψεις τους, ώστε να εξευρίσκονται στη συνέχεια λύσεις στα προβλήματα επί τόπου. Διότι γνωρίζουμε ότι η πολιτική συνοχή αφορά την εσωτερική συνάφεια και συνοχή των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να προωθεί και προαγάγει την περιφερειακή ανάπτυξη και πρέπει να βοηθήσουμε οι κοινωνικές στενοποί και τα κοινωνικά προβλήματα να διεκπεραιώνονται και να επιλύονται. Τα προβλήματα αυτά πρέπει να τη χάνουν αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε με αλληλέγγυο τρόπο να αντιμετωπίζονται. Είχαμε και την αντίφαση, η αντίθεση ότι στις περιφέρειες μας έλεγαν ότι θα έπρεπε να καταβάλουμε προσπάθειες στις διατάξεις και τον κανονισμό να μην είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στην θεματολογική επικέντρωση θεματολογική επικέντρωση όσον αφορά για παράδειγμα αριθμό και πλαίσια σχεδίων αλλά οι ανάγκες που είναι διαφορετικές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση των λειτουργικών προγραμμάτων ώστε να υπάρχει ελαστικότητα και να μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Από την άλλη πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εσά, η θεματολογική επικέντρωση ετίθετο πάντα στο επίκεντρο και μάλιστα με το σκεπτικό ότι τα κονδύλια τα οποία θα επιμεριστούν, τα χρήματα που θα μοιραστούν θα είναι λιγότερα πλέον. Και με αυτά τα επιχειρήματα, λιγότερα λέει χρήματα θα έχουμε και πρέπει να επικεντρωθούμε θεματολογικά σε, συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένους άξονες για τους υπεύθυνους ε, για αυτά τα προγράμματα η διαβούλευση αυτή αποκλείεται και λένε ορίστε έχουμε δύο-τρία κέντρα βάρους. Αυτά ούτως ή άλλως τα θέλαμε να υπάρχουν. Ε, αυτά θα υλοποιηθούν τώρα με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Όμως αυτό δεν είναι το νόημα και το σκηνικό για αυτή την πολιτική για την περιφερειακή ανάπτυξη. Αν συνεχιστούν τα πράγματα όσο έχουν τώρα, αυτά τα οποία σε 10-15 χρόνια και χώρες που είναι για μεγαλύτερο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φορείς ευρωπαϊκών σχεδίων και προγραμμάτων, Τώρα τι θα γίνει. Θα παραμείνουν αυτοί εκτός και δεν θα μπορούν να συμπεριληφθούν στη διαδικασία διαμόρφωσης και κατάτησης των προγραμμάτων. Θα έπρεπε να αποφύγουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ. το Για όλο το θέμα της ευρυζωνικής σύνδεσης. Είναι ένα θέμα που έχουμε σε κάποιες χώρες. Ουσιαστικά τι συμβαίνει. <clears throat> Περαιτέρω επενδύσεις πρέπει να γίνουν πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κονδύλια των διαθροτικών ταμείων για παράδειγμα. Όπως όταν υπάρχει μια αριθμία ή ένα πρόβλημα της αγοράς, όταν για παράδειγμα δεν μπορεί κάτι να είναι αποτελεσματικό και κερδοφόρο σε μια αγορά, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η δράση, πρέπει να διασφαλιστούν αυτές οι επενδύσεις. Με τους συναδέλφους μας από πλευράς Άγκρη βρισκόμαστε σε συζήτηση για αυτά, διότι πιστεύουμε ότι στον χώρο της υπαίθρου πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη και το πρίσμα της περιφερικής ανάπτυξης, πράγμα το οποίο συνεπάγεται και την χρήση μεγάλων, πολλών κονδυλίων και αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε μπορούμε να το συμμεριστούμε ως έργο. Από περίπτωση αναπερίπτωση πρέπει να εξετάζουμε και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Έχουμε 7 χώρες όπου αυτό θέτει ένα ζήτημα. Στη Γερμανία υπάρχουν κάποιες περιφέρειες της πρώην Ανατολικής Γερμανίας οι περισσότερες και μία περιφέρεια στην πρώην Δυτική Γερμανία. Πρέπει αναπερίπτωση να δούμε ποια απόφαση μπορεί να ληφθεί. Δεν αποκλείεται να μπορεί να γίνει αυτό, αλλά πρώτον πρέπει ακριβώς να δούμε σε τι οφείλεται μια αποτυχία ή αριθμία της αγοράς. Δεύτερον, να δούμε τι πρέπει πρώτα να γίνει. Δεύτερον, και να δούμε η ιεράρχηση και προτεραιοτήτων μέσα στο πλαίσιο αυτού του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Να δούμε τι πρέπει πρωταρχικά να γίνει ώστε όταν πρόκειται για το χώρο της υπαίθρου να μπορούμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου να συνεισφέρουμε με αυτές τις δράσεις. Ως προς αυτό διεξάγονται αντίστοιχα συζητήσεις και διαβουλεύσεις για το όλο το θέμα των εταιρικών σχέσεων έχετε μια αισιόδοξη προσέγγιση είπατε και είναι σωστή, σωστή αυτή η προσέγγιση. Αν τώρα μια χώρα κάποιες εβδομάδες πιο πριν ή κάποιες εβδομάδες με κάποια καθυστέρηση θα προχωρούσε, δεν είναι αυτό το αποφασιστικό στοιχείο. Υπάρχουν αποφάσεις που πρέπει να ενταχθούν και να λαμβάνονται υπόψη και να συμμορφωνόμαστε με αυτές. Το μεγαλύτερο τμήμα των συζητήσεων <clears throat> θεμελιώνονται σε σχέση με τα κράτη-μέλη, βασίζονται σε θέματα που ήδη πέρι, ε, το, κατά τα μέσα ε, του θέρους ε, έχουν ρυθμιστεί για το τι πρέπει να γίνει, ποιες καινοτομίες ή τροποποιήσεις και αλλαγές θα, θα συνεπάγονται σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων. Αυτή είναι η θεματολογική επικέντρωση. Αυτή είναι στοχοθέτηση, στοχοπροσύλωση όσον αφορά τις πολιτικές μας και η υλοποίηση των εξάντε όρων και προϋποθέσεων, των εκπροημίου όρων και προϋποθέσεων. Η κατάθεση στρατηγικής στρατηγικών, για παράδειγμα market specialization, εξειδίκευση για την, στην αγορά, μεταφορές. Υπάρχουν λοιπόν ανάπτυξη, στόχοι ανάπτυξης με βάση στρατηγικές και όχι το αντίστροφο, στρατηγικές με ανάπτυξη. Λοιπόν, πρέπει να δούμε το ευρύτερο πλαίσιο, τη σφαιρική εικόνα. Είναι μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έχουμε τώρα, ότι στους πιο διαφορετικούς τομείς τι συμβαίνει έχουμε υποβολή ε, στρατηγικών που θα κατατίθενται, που θα εξηγούν και θα αποδεικνύουν γιατί και πώς θα πρέπει να γίνονται κάποιες επενδύσεις και με ποιο στόχο. Σε κάποιες ε, χώρες μέλη έχουμε ε, στόχο να επενδύσουν τα κράτη στον τομέα υγείας. Ε, δεν είναι αυτό η πρώτη μας προτεραιότητα. Μπορούμε να πούμε εντάξει, βαίνει καλό αυτό, μπορεί να γίνει, όταν υπάρχουν επαρκώς αιτιολογημένα σχέδια γιατί πρέπει να γίνουν τέτοιες επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Αυτό είναι μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και είναι ας το πω έτσι πρόσθετη προσπάθεια που απαιτείται από αυτά. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό και για τις υπηρεσίες μας απαιτείται πρόσθετη προσπάθεια. Πρέπει να συλλέξουμε πείρα αρκετή για να προχωρήσουμε καλά. Μέχρι τα τέλη Απριλίου όμως αυτές οι εταιρικέ σχέσεις, αυτά τα, οι συμφωνίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν ολοκληρωθούν με αναγκαία στοιχεία και ανταλλαγή στοιχείων. Για την Κροατία το ανέφερα ήδη το πρόβλημα που υπάρχει, ώστε όλοι να μπορούν να τηρούν τα αναγκαία στοιχεία μέσα στα αναγκαία πλαίσια. Και πώς να το πω, τα πιο εξειδικευμένα σχέδια και προγράμματα που αφορούν εσωτερικές διαβουλεύσεις και ε, διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να μπορούν να επιταχυνθούν ώστε στο τέλος τα περισσότερα προγράμματα να μπορούν μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο, χρονικό πλαίσιο, χρονοπλαίσιο να εγκριθούν και να προχωρήσουν. Εξακολουθώ να πιστεύω μέσα στη σημερινή συγκυρία ότι από ένα εξάμεινο μέχρι ενός έτους θα πρέπει να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ε, βελτιωμένα σε σχέση με πέρυσι. Εφέτος και του χρόνου, το 2014, το 2015 η ε, εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων με βάση τα πραγματικά σχέδια και στόχους θα πρέπει να βρεθούν στο προσκήνιο της τα πραγματικά επιτεύγματα. Και έτσι με τα νέα προγράμματα που θα κατατεθούν, όταν πρόκειται για προγράμματα για τις υποδομές, έχουμε την κατάσταση σε κάποιες, κάποιες χώρες ότι πρέπει να ξεχωριστούν, να διαχωριστούν αυτά τα προγράμματα και σχέδια από τη μία περίοδο προς την άλλη. Να γεφυροποιηθεί η δυνατότητα συνέχισης με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων από τη μία περίοδο στην άλλη. Δεν έχω καμιά ανησυχία βέβαια ότι θα μπορέσουν να να καλυφθούν οι ανάγκες και να συνεχιστούν αυτά τα προγράμματα. Αυτά είναι τα ουσιοδέστερα και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο υπό τη δική μου προσέγγιση θέλω να πιέσω να προχωρήσουμε ταχύτερα. Ιδιαίτερα οι επενδυτές στον ιδιωτικό τομέα να έχουν προσανατολισμούς και κατευθυντήριες γραμμές τι σε ποιου τομεί θα είναι διαθέσιμο και διαθέσιμα ώστε να μπορούν να κάνουν το σχεδιασμό τους και τον προγραμματισμό τους έγκαιρα και αποτελεσματικά. Αυτό είναι το αποτελεσματική σημασία στοιχείο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήδη σήμερα μπορούν τα κράτη-μέλη να καταθέτουν ε, σχέδια και να προχωρούν και να συγχρηματοδοτούνται όταν ταιριάζουν αυτά τα σχέδια αυτών των προγραμμάτων στο δικό μας, στις δικές μας αρχές. Και έτσι όταν μπορούν με αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο να εγκριθούν. Τώρα, προγράμματα για τον πολιτισμό. Όταν συνεισφέρουν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης με αηφόρο βιώσιμο τρόπο, θα αποτελούν τμήμα των κανονικών πολιτικών μας και διαδικασιών μας. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη εναντί των άλλων δραστηριοτήτων. Αυτό για κάποιες χώρες έχει μεγάλη σημασία σήμερα θα έλπιζα αυτή η εμβέλεια, αυτή η σπουδαιότητα να αυξηθεί για πολλές χώρες, ώστε ένας αυξανόμενος αριθμός των εμπλεκόμενων στην αγορά, σε ένα σημαντικό τομέα στην Ευρώπη, στον τομέα αυτόν για την Ευρώπη, που έχει σημαντικό δυναμικό, να μπορέσει να αναπτυχθεί. Κύριε Όλμπρεχτ, δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αντίθεση ε, σε σχέση με τις delegated acts, τις κατεξουσιοδότηση πράξης ε, όσον αφορά τον αριθμό για παράδειγμα θεμάτων που θεματολογικά μπορούν να διεκπεραιώνονται μέσα από μια τέτοια πράξη. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κατεξουσιοδότηση πράξη ή να υπάρχει ένα πακέτο μέτρων μέσα σε μια τέτοια πράξη, ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Υπάρχει ανάγκη πολλές φορές να συζητηθούν κάποια πράγματα και να διευθετηθούν. Ελπίζω ότι αυτά δεν θα οδηγήσουν όμως σε καθυστερήσεις. Ελπίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα. Ξέχασα τίποτα. Όχι, δεν ε, τελειώσαμε γιατί ακόμη έχουμε άλλους τρεις που μας τις το uh, Καλά, εάν τα έχετε απαντήσει με καλύψει, θα σας το πούνε. Κύριε Χρυσόγελε. Ε, ακούω προσεκτικά αυτό που είπατε και για τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά πώς αντιλαμβάνονται ένα βασικό στοιχείο ε, της νέας προγραμματικής περίοδου που είναι το bottom-up approach. Δηλαδή, την ουσιαστική διαβούλευση πρέπει να γίνει στο πλαίσιο κάθε περιφέρειας, όχι μόνο με τον Περιφερειάρχη, τις Περιφερειακές Αρχές, αλλά με την κοινωνία των πολιτών. Νομίζω ότι επειδή ακριβώ υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις και εγώ βλέπω ότι αντιλαμβάνεται αυτό το διάλογο σαν μια ημερίδα όπου διάφοροι φορείς έρχονται και μιλάνε και θεωρούν ότι εκπληρώθηκε η προϋπόθεση της επόμενης προγραμματικής περίοδου και για να μην υπάρξουν εκπλήξεις θα περίμενα και από την Κομισιόν λίγο να φτιάξει ένα οδηγό τι είναι και τι δεν είναι ουσιαστική διαβούλευση, αυτή το bottom-up approach. Για να μην έρχονται εκ των υστέρων τα κράτη-μέλη ή περιφέρειες και να λένε «Μα δεν το είχαμε καταλάβει». Το, δεύτερο είναι αυτή η θεματική προτεραιότητα που είναι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το θέμα της έρευνας, τεχνολογίας και μέσω της εφίους εξειδίκευσης. Και υπάρχει υποχρέωση για να χρηματοδοθούν αυτές οι δράσεις να υπάρξει σχέδιο στρατηγικής, να υπάρχει στρατηγική καταρχή και να υπάρχει και ένα σχέδιο δράσης το οποίο πάλι θα πρέπει να προκύψει μέσα από ουσιαστική διαβούλευση. Πάλι φοβάμαι ότι αυτές οι περιφέρειες που έχουν εμπειρία ήδη από παλιά μπορούν να το υλοποιήσουν αυτό, αλλά δεν έχουν καταλάβει αν οι περιφέρειες αντιλαμβάνονται, οι άλλες περιφέρειες που δεν έχουν αυτή την εμπειρία, έχουν ενημερωθεί συστηματικά. Και εκεί, και όπως είπε και ο συνάλφος, νομίζω ότι χρειάζεται μια απεύθυνση όχι μόνο στο κράτος μέλος ή στις περιφερειακές αρχές, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία, σε μερικά βασικά κομβικά θέματα της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Δηλαδή, να μην συγχαίνω ότι η έρευνα είναι μόνο το Horizon 2020 ή να μην θεωρούν ότι απλώς γίνεται στην περιφέρεια μία μελέτη, την υιοθετεί η περιφέρεια και αυτό ήτανε. Ε, ε, είναι πολύ διαφορετικέ οι προσεγγίσει νέα περίοδου. Μέχρι τώρα όμω σκεφτόταν με το άλλο μοντέλο, ενώ τώρα αλλάζει. Και δεν είμαι σίγουρο ότι όλε οι περιφέρειες έχουν καταλάβει καταρχή κάτι τέτοιο. Ε, ένα τρίτο θέμα που αφορά τη μεταφορά σε πολλές περιφέρειες έχει γίνει το λεγόμενο overbooking. Δηλαδή έχουν εντάξει πολλά προγράμματα μέσα με αποτέλεσμα ο προπολογισμό να είναι 130% σε σχέση με το πρόγραμμα που τρέχει 2007-2013 και κάποια έργα δεν θα τελειώσουν. Επομένως, ή θα πιέζουν να μεταφερθούν τα έργα αυτά στην επόμενη περίοδο, που όμως δεν εντάσσονται στρατηγική αυτή που έχουμε αφασίσει για τους κανονισμούς της επόμενης περίοδου, ή θα πρέπει να επιστρέφουν χρήματα, γιατί τα έργα αυτά δεν θα είναι επιλέξιμα. Πώς θα έχετε αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι πάρα πολλές περιφέρειες πιέζουν ένα 20-30% 40-50% είναι μεταφορά έργων από την προηγούμενη περίοδο στην επόμενη. Ε, και ένα τελευταίο είναι, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα σε χώρες της κρίση που είναι και στο πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αναφέρθηκε και από άλλους, ε, η εθνική συμμετοχή είναι δύσκολη, δεν ξέρω αν θα δεχόνταν η Κομισιόν να θεωρήσει ότι η συνεισφορά των κρατών μελών αφαιρείται από, τους, από, τα, δημο, ε, τις δημόσιες δαπάνες και άρα δεν υπολογίζεται στο έλλειμμα. Γιατί από ό,τι θυμάμαι αυτό είχε απορριφθεί και στη δικιά μας επιτροπή και εγώ το είχα καταθέσει αν θυμάμαι καλά ως τροπολίγια αλλά αυτό είχε απορριφθεί. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να δεχτεί κάτι τέτοιο, δηλαδή ότι η εθνική συμμετοχή στα έργα δεν υπολογίζεται τελικά στο έλλειμμα. Και αυτό θα ήταν μια σημαντική πληροφορία για τα κράτη-μέλη. Και το δεύτερο είναι ότι σε ορισμένες χώρες τα, μέσα στα εναλλακτικά ε, συστήματα χρηματοδότηση μακροοικονομικά, όπως ψηφίσαμε και εμείς εδώ, είναι το θέμα των συνεταιριστικών τραπεζών. Σε μερικές χώρες υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, στην Αυστρία, στη Γερμανία, ε, Γαλλία και...